Varmt välkomna och vi återupptar. Καλημέρα σας. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Σήμερα έχουμε τις ε, ψηφοφορίες και θα πρέπει να συζητήσουμε με την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ. Και θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε και ένα σωρό άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο σημείο είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα. Είναι το σημείο 11. Και θα περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Για το σημείο 11. ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα ήτρε. Θα ψηφίσουμε unblock από την τροπολογία 4 στο 3 unblock υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και μετά τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ την κυρία Τόμσεν ε, για τις τροπολογίες της. Σημείο 12. Πώς θα αυξηθεί ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίζουμε, Ψηφίζουμε κατευθείαν τρόπολογια υπερθμών 3 ψήφι υπέρ κατά απόχες ενεκρίθησαν. Τροπολογία 4. Θα κάνουμε έλεγχο. 4. Άρχεται. Ναι, ναι, τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Uh, 12-13. Απορρίπτεται. ο um, Πρόεδρε, ξέχασα την κάρτα μου και ο βοηθός μου έρχεται. Μπορείτε να σημειώσετε ότι καταψήφισα. Υπέρ, λέει Κατά αποχές. Ελέγχουμε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 4 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 5 με 1. Ψηφίζουμε από, κοινού, από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτές. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιαρόκοα για να προεδρεύσει. morning, and Καλημέρα σας. Καταρχήν εκφράζω την χαρά μου που ψηφίζουμε την ε, έκθεση της Προέδρου μας με τη βοήθειά μας. Με τη βοήθειά μου θα προσπαθήσω να το κάνω στο δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Μήπως μπορώ να σας δώσω το λόγο κυρία Πρόεδρε και η εισηγήτρια. Θα είμαι πολύ σύντομη. Εγώ ήθελα απλώς να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους και όλη την Επιτροπή, διότι βλέπω ότι πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ θέληση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο όσο το δυνατόν καλύτερο. Προσπάθησα να συγκεντρωθώ σε αυτό το που είναι πραγματικά ουσιαστικό για να μην συντάξω ένα μακροσκελές κείμενο. Θέλησα να είμαι πολύ συγκεκριμένη σε αυτά που προτείνουμε. Επίσης, ε, δέχτηκα και πολλές από τις ε, τροπολογίες οι οποίες αποτελούν βελτίωση για το κείμενο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία συγκεκριμένη έκθεση, σαφή έκθεση, χωρίς να έχουμε ένα φλίαρο κείμενο, Ήθελα ακριβώς να είμαι σαφής στις προτάσεις μας. Απέσυρα και εγώ αρκετές τροπολογίες μου για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πυκνό κείμενο. Και ελπίζω ότι θα υποστηριχθεί ευρέως από την, Κομισιό, από την Επιτροπή μας διότι πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό για την ισότητα των φύλων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Εισηγήτρια και ξεκινάμε με τους συμβιβασμούς. Έξι Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ένα, Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεκτή. Συμβαστική δύο, Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 57 υπέρ <clears throat> κατά αποχές απορρίφεται. Ή αν θέλετε να ελέγξουμε για την 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Δεκατρεις υπέρ. Τροπολογία 58 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίφονται. 60 υπέρ κατά. Μόνο αν η 58 είχε εγκριθεί θα είχε εκπέσει 60. 60 ψήφι υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 ψήφι υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά. πρέπει να έλεγξουν. Έλεγχος ηλεκτρονικός στην 61. Πέρας, ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ, 1 κατά. 10 αποχές. 62 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 63. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ Α, εκπίπτει, συγγνώμη. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 69 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί και αυτή. 69 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές Μήπως μπορούμε να την ελέγξουμε, την 70 παρακαλώ. Πέρας 70 απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά Αποχές. <clears throat> Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Α το ελέγξουμε όμως. Τροπολογία μόνο 80. Και την ψηφοφορία. Πέρασε. Πράγματι απέριπτε. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 81 έχει εκπέσει 70. Μα δεν είναι κριτή 80, κυρία Πρόεδρε. Α, συγγνώμη, 81, μεγάλο το δίκιο σας. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. Ας ελέγξουμε. Αρχή την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. εκπίπτει 78. Πάμε στο 83. 82 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Με μία ψηφοδιαφορά διαφορά απερίφθη. Ενενήντα ψήφοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 Ας ελέγξουμε την 90 προηγουμένως. Έλεγχος την 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται όπως έλεγα 18-15. Μάλιστα. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Πάτησα κατά ενώ έπρεπε να πατήσω υπέρ. Συγγνώμη, υπέρ. Και πάλι απορρίπτεται, κυρία μου. Κυρία Φιγκερέιντου, και εγώ έκανα λάθος, πάτησα άλλο, πάτησα άλλο κουμπί και συνέβη σε μένα το ίδιο και με την κυρία Κώστα. Μήπως θέλετε να επαναλάβετε την ψηφοφορία. Πάλι απορρίπτεται 17-18 λέει η πρόεδρος. Ας ξαναψηφίσουμε 87 άθετη ψηφοφορία. Η 90, συγγνώμη. 90. 9-0. Ψηφίσουμε την 90. Την 90 Τροπολογία 90 άρχεται πέρας ψηφοφορία. 17-16, όπως το προέβλεψε ο κύριος Ταραμπέλα που ξέρει μαθηματικά. Η 87 εκπίπτει, η 86 εκπίπτει, η 88 εκπίπτει, 89. Ψήφι υπέρ, κατά αποχές Δεν ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της ίδιας. Τροπολογία 91. 91 είπα. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. <clears throat> Δεκτή. 92 Εκπίπτη. 93 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95. Έλεγχος για την 93. Αρχιτεί ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 με 21. 96 άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 97 υπέρ. 97 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 μποσκούρτ ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 101 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή 103 υπέρ κατά αποχές απορρίβεται έλεγχος για την 103 άρχεται πέρασε απερίφθη 105. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140 τμήμα τμήμα 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 140 τμήμα 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 106 έχει αποσυρθεί. Εκατόν 114 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 114. Πέρας. 19-13 εγκρίνεται πράγματι, συγγνώμη. Γλωσσικού χαρακτήρα είναι η επόμενη, δεν την ψηφίζουμε. Και περνάμε στην 108. Εκπίπτει και 112 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Ναι, έλεγχος. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία για την 113. Εκατόν δεκατρία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 117 θα ψηφιστεί αργότερα. Πάμε στην... Πάμε στην 120 της κυρίας Χάνιμπολ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές ας την ελέγξουμε 127 αρχιτή ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται 14 18 κατά. Το 23 και 125 <clears throat> ψηφιπέ κατά. Αποχές απορρίπτονται. Εκατόν ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά ας ελέγξουμε. Καλού κακού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται 17-15. Καλά που ελέγξαμε. 128 με, σε τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι πέρα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. <clears throat> Κατά αποχές απορρίπτεται. 1.29 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, <clears throat> τουλάχιστον έτσι νομίζω, ας, ας ελέγξουμε. 129. Άρχεται η ψηφοφορία, λέει. Πέρας. 15 υπέρ 16 κατά απερίφθη. 131 ψήφι υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 132 εκπίπτει, 133 αργότερα, 134 ψήφι υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 1.35 υπέρ, κατά, εποχές δεκτή, 136 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός για την 136. Πέρας. 15 υπέρ 16 κατά απορρίπτεται. 137 είναι η επόμενη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Λοιπόν, 137, σηκώστε πάλι Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 1, 3, 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στην 142. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές δεκτή 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 147 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 13 υπέρ, 19 κατά απορρίπτεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές Ας το ξανακάνουμε με χέρια, όχι ηλεκτρονικά. 151. Ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εν, εν, απορρίπτεται. 155 εγκρίνεται πράγματι, αλλά ας την ελέγξουμε. στις προφορίες. Εγκρίνεται, εγκρίνεται σαφώς με ένα. Ναι. εγκρίνεται λοιπόν. 156 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν... 154. Ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 157. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 160. Υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. 160. Πέρας, ψηφοφορίες. Okay. So it is... Εγκρίνεται, μάλιστα. Η επόμενη είναι η 168 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος, επαλήθευση. Για την 168, άρχιτε ψηφοφορία, 168. Πέρας ψηφοφορίας, 32 ψήφισαν, 15 υπέρ 16 κατά. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές Επίσης απορρίπτεται 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 163 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 164 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100... Ε, επαλήθευση για την 166 ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Σχεδόν. Ναι, απορρίπτεται. Με διαφορά τέσσερων ψήφων. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 172 καταπίπτει... Καταπίπτουν όλες μέχρι την 176 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ ε, η 175 διορθώνει η πρόεδρος υπέρ 175 κατά αποχές επαλήθευση για την 175 παρακαλώ πέρας Απορρίπτεται με διαφορά τριών ψήφων. 177 καταπίπτει. 178 Ψηφίζουμε για την 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. 179 καταπίπτει. Κυρία Τόμψεν, θέλετε παλήθευση. 178 τότε, ξαναψηφίζουμε. Παρακαλώ. Πέρας. Η ισοψηφία απορρίπτεται. 180 τώρα. Εκατόν ογδόντα υπέρ κατά αποχές Κατόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 183 ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 22 προς 9 και μία αποχή. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, επαλήθευση για την 9 παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας όχι ακόμα. πέρα τώρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Υπέρ για την 8. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτουν ε, οι επόμενες. Οι 11, οι 15 και οι 14, 12 τώρα υπέρ. 12. Τροπολογία 12. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι 16 καταπίπτει. 13, 19, στη 18 φτάνουμε τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση παρακαλώ για την ε, τροπολογία 18. Πέρας της ε, ψηφοφορίας απορρίπτεται όντως. Η τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 καταπίπτει. Θα ψηφίσουμε για την 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 27 ήταν ταυτόσημη με την 24. 23 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση παρακαλώ για την 30 πέρας ψηφοφορίας ναι απορρίπτεται 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση για την 34 σας παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 15 υπέρ 16 κατά μία αποχή απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, ε, επαλήθευση παρακαλώ για την 38. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 38. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41. Κατά τμήματα ψηφοφορία το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 41 παρακαλώ. Πέρας. Ναι, εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Η 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές. 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 40, Ε, πάλι δεν αν θέλετε. Ποιο ζήτησε κανένας. Καταπίπτει 46... 45. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Α το ελέγξουμε. Για τη 45 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία. 15 προς 14 ε, είναι η ψήφη, εγκρίνεται. 47 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ορίτε. 48 Υπέρ. Στι 48 έχουμε φτάσει. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 49 καταπίπτει ή 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση για την 53 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Πέρας. Για την 54 πάντοτε έτσι. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε. Ελπίζω να μην χρειαστούν άλλοι έλεγχοι. 56 ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται 18 προς 11. Ας περάσουμε στην αιτιολογική σκέψη. Τροπολογία είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 4 τώρα υπέρ κατά άποχες επαλήθευση γιατί δεν με προλάβατε βλέπω Τέσσερα. ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τέσσερα, παρακαλώ Απορρίπτεται, έχουμε ισοψηφία. Τροπολογία 5 κατά αποχές Πορύπτεται. τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τέλος τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται και τώρα θα προβούμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Φένσον. People won. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. And it's adopted with 27. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ καμία κατά δύο εποχές συγχαρητήρια. Just Προς ενημέρωσή σας, θα αρχίσουμε λίγαν συντόμως, αναμένουμε την Επίτροπο Ρέντινγκ. Ε, υπομονή, λίγα λεπτάκια. Κυρία Σινκλέρ, ε, εφόσον περιμένουμε θα ήθελα να πω κάτι. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε την Διεθνή ημέρα των γυναικών και είχαμε ένα πρόγευμα με τον πρόεδρο Μπαρόσο και την αντιπρόεδρο Ρέντινγκ. Το έχω ξαναπεί στην Επιτροπή και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ε, κυρία Σβένσον, εφόσον είστε γυναίκα ποιότητας. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να παρευρεθούμε σε τέτοιες συναντήσεις. Ξέρω ποια είναι η επίσημη απάντηση. Ε, αλλά πώς αυτό αποκαλούνται όλοι οι δημοκράτες ε, όταν εκπροσωπ... κάποιοι εκπροσωπούν 5 εκατομμύρια ανθρώπους και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να του εκπροσωπήσουν γιατί η χώρα του ολόκληρη δεν έχει πληθυσμό 5 ε, εκατομμύρια. Συγγνώμη, αλλά ε, ε, στη... εγώ πηγαίνω, στη... δεν μπορώ να έρθω στη συνεδριάση συντονιστών, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την ψήφο μου για να διορίσω κάποιον. Γιατί μου αρνείστε τη συμμετοχή στη συνεδρίαση των συντονιστών, γιατί δεν έχω ισότιμη μεταχείριση. Πρόεδρος. Ε, ευχαριστούμε που θίξατε αυτό το ζήτημα και να διευκρινίσουμε περί τίνος πρόκειται. Πρώτον, Υπάρχει ένας κανόνας που δεν ισχύει μόνο για την Επιτροπή μας, αλλά ισχύει για όλες τις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και για την ε, Διεθνή ημέρα γυναικών τη συνέβη. Ήταν προσκεκλημένοι συντονιστές της Επιτροπής από τον πρόεδρο Μπαρόσο. Οι συντονιστές δυνάμει αυτού του κανονισμού προσκαλούνται. Και στην προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος Μπαρόσο είχε απευθύνει την πρόσκληση προς τους συντονιστές. Είναι ένας κανόνας καθιερωμένος που σας λέω διέπει τις εργασίες όλων των επιτροπών. Ε, δεν μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε, να τροποποιήσουμε αυτόν τον κανόνα. Θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση να τροποποιηθεί ο κανονισμός. Εμείς ως Επιτροπή πάντως δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα η κυρία Σινκλέρ επερώτηση. Ήρθε η Επίτροπος Ρέντινγκ και θα ήθελα να ακούσει για τι πράγμα συζητάμε. Έλεγα για το πρόγραμμα της περασμένης εβδομάδας ε, όπου δεν μπόρεσα να παρευρεθώ γιατί δεν είμαι συντονίστρια. Λέτε, ε, πρόεδρε δεν μπορείτε να επηρεάσετε τους κανόνες άμεσα. Όχι, ε, συμφωνώ, αλλά μπορείτε να ζητήσετε εκπροσώπηση της Επιτροπής. Θα ήθελα κάποιο χρόνο αγόρευσης, κάποια εκπροσώπηση ε, νομίζω ότι αυτό εντάσσεται στην εντολή που έχετε ως Πρόεδρος και θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξη από συναδέλφους. Αν, αν κάποιοι δεν ε, υποστηρίζουν τη συμμετοχή μου στις δημοκρατικές διαδικασίες του Κοινοβουλίου θα ήθελα να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν με υποστηρίζουν Πρόεδρος. Όπως σας είπα και ε, προηγουμένως, είναι ένας γενικός κανόνας αυτός ε, που ισχύει για όλες τις επιτροπές. Αν ζητάτε κάτι συγκεκριμένο, κυρία Σίνκλερ, μία ερώτηση έκανα, πρόεδρε, διακόπτε, κυρία Σίνκλερ. Απάντησα αυτή την ερώτηση και μπορώ να σας πω το εξής. Είναι γενικό ο κανόνας, δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε ω Επιτροπή αυτόν τον κανόνα. Αν όμω το επιθυμεί η κυρία Σινκλέρ, ε, μπορώ στη διάσκεψη των Προέδρων όπου είμαι μέλος να υποβάλω το ερώτημά σας κυρία Σινκλέρ. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Σας ικανοποιεί. Μάλιστα. Φτάσαμε στο σημείο 14 της ημερησίας διατάξεως. Σας καλωσορίζουμε θερμά, κυρία Ρέντινγκ. Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε τις ε, προτεραιότητες στην Επιτροπή και προσβλέπουμε σε οποιαδήποτε ενημέρωση μπορείτε να μας δώσετε για τα θέματα άμεσα αρμοδιότητας Επιτροπής μας, τα θέματα ισότητας των δύο φίλων. Σας καλωσορίζουμε θερμά και θα σας δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο. Έχουμε στη διάθεσή μας μια μισή ώρα για την ε, ανταλλαγή απόψεων και για τη συζήτηση. Ευελπιστώ ότι σε αυτό το διάστημα, το οποίο ελπίζω να τηρήσουμε, Ελπίζω λοιπόν να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλώς ορίσατε και πάλι και σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχαμε συναντηθεί με ορισμένες από εσά τουλάχιστον πρόσφατα και να είμαστε πάλι εδώ. Έχουμε μια επίσημη ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας την ισότητα των φύλων. Θέλω καταρχήν να σας πω <clears throat> πόσο χαιρετίζω την έκθεση της ε, Μαρία Νιδέλτσεβα και της Ιωάννα Πλαμπ για τα θέματα ισότητας και ένδυας που ενεκρίθη την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Πρόκειται για σημαντικά στοιχεία τα οποία φυσικά θα λάβουμε και υπόψη μας στο έργο μας γνωρίζετε ότι η ισότητα των φύλων παραμένει ένας στόχος ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί. Δυστυχώς παραμένουν ακόμα σημαντικές ανισότητες. Οι γυναίκες ε, εργάζονται σε ίσες συνθήκες, αλλά πληρώνονται λιγότερο από τους άνδρες και δεν εκπροσωπούνται όσο θα έπρεπε να εκπροσωπούνται σε θέσεις όπου μπορούν να είναι υπεύθυνε για τη λήψη αποφάσεων. Αν μπορώ τώρα να κάνω μια επισκόπηση του τι έχει γίνει από πέρσι μέχρι τώρα. <clears throat> Καταρχήν πέρσι ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την ισότητα των φίλων, γιατί για πρώτη φορά η Κομισιόν ανέλαβε τη δέσμευση να εισαχθεί η ισότητα των φίλων σε όλο το πολιτικό της έργο. Ήταν μια χάρτα για τις γυναίκες που ο πρόεδρος της Κομισιόν και οι υπόλοιποι επίτροποι προσυπέγραψαν και ακολουθήθηκε από τη διατύπωση μιας στρατηγικής για την ισότητα ανδρών και γυναικών στις 21 Σεπτεμβρίου του 2010 και του σχεδίου δράσης για την προώθηση της ισότητας αυτής μεταξύ 2010 και 2015. Έχουμε λοιπόν πραγματικά ένα οδικό χάρτη περί του πρακτέου στα επόμενα χρόνια για την επίτευξη αυτής της ισότητας. Θυμάστε ποιε ήταν οι πέντε προτεραιότητε. Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι η πρώτη. Και εδώ μπορώ ήδη να σας καταδείξω πως η χάρτα είχε κάποια επιρροή στην διαμόρφωση της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, γιατί πράγματι ελήφθησαν υπόψη τα θέματα των γυναικών σε πολλά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη το ποσοστό από απασχολησιμότητας του 75% για την Ευρώπη του 2020, ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μονάχα εάν χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό των γυναικών, το οποίο μέχρι στιγμής είναι ανεκμετάλλευτο. Και αν βελτιώσουμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Επομένως, η ισότητα των φύλων είναι και ένας σημαντικός πυλώνας των κατευθυντηριών γραμμών για την απασχόληση. Επίσης, <clears throat> το θέμα της ανισότητας εισοδημάτων. Γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η διαφορά. Υπάρχει το υψηλό ποσοστό της ατυπικής εργασίας των γυναικών και επίσης οι διακοπές καριέρας που οδηγούν σε ένα μέσο όρο ο οποίος είναι χαμηλότερος για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες και φυσικά αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ένδια των γυναικών, σε χαμηλότερες συντάξεις για τις γυναίκες και στον κίνδυνο να υπάρξει ένδια σε μεγάλη ηλικία για τις γυναίκες. Και εξάλλου η Κομισιόν σχεδιάζει να εκδώσει μια λευκή βίβλο για τις συντάξεις το 3ο 4 ο του 2011 και εδώ και πάλι το δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων και την κοινωνική συμπερίληψη θα συμμετάσχουν στο έργο αυτό. Θα, θα δείξει λοιπόν αυτό και πάλι την επιρροή της χάρτας για την ισότητα. Σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλουν οι συναδελφοί μου λοιπόν λαμβάνουν υπόψη τη χάρτα για την ισότητα των φύλων. Ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο βέβαια είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξή σας, είναι η συμφιλίωση τη επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ξέρουμε όλοι ότι οι στόχοι της Βαρκελόνης για την παιδική φροντίδα δεν έχουν επιτευχθεί. Τουλάχιστον για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν επιτευχθεί και στις υπόλοιπες όχι στο επίπεδο που θα θέλαμε να έχουν επιτευχθεί και τα κράτη-μέλη επομένως θα πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Άψκο κατεγράφει αυτό Είπαν οι υπουργοί, βεβαίω έχουμε στόχου, συμφωνούμε με του στόχου και μετά δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν, ότι οι στόχοι τη Βαρκελόνη για την παιδική φροντίδα δεν έχουν υλοποιηθεί. Το θέμα της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής περιλαμβάνει επίση το θέμα της μητρικής άδεια, της οδηγίας για τη μητρική άδεια. Ξέρετε ότι αυτή η οδηγία είναι μπλοκαρισμένη <clears throat> γιατί η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση θεωρείται από το Συμβούλιο ή τουλάχιστον από πολλές χώρες μέλη ως απαράδεκτη και επομένως αρνούνται κάτι κατηγορηματικά να συζητήσουν το θέμα αυτό, το έχουν βάλει στο ράφι και απλώς το κάνουν αυτό για να δείξουν ότι είναι ενοχλημένες από τη θέση του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό εγώ πήρα την πρωτοβουλία, κυρία Πρόεδρε, χωρίς καν να ζητήσω την ε, άδειά σα να συζητήσω με τις επερχόμενες προεδρίες και να δούμε αν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το αδιέξοδο. Γιατί όλοι παραμένουν στη θέση τους χωρίς μετακίνηση. Αυτό όμως δεν ωφελεί εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση. Γιατί να μην επανέλθουμε λοιπόν στο κείμενο της Κομισιόν, το οποίο φυγραμμίζεται με τα πρότυπα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, και δεν επιβάλλει ένα δυσβάστακτο κόστος στα κρατημέλη μελη σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό τους, που είναι φυσικά προϋπολογισμός λιτότητος ήδη. Ίσως λοιπόν το κείμενο της Κομισιόν θα μπορούσε να αποτελέσει βάση συμβιβασμού και θέλω εδώ να προσθέσω και μια πολύ καλή ιδέα η οποία περιλαμβανόταν στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η ρήτρα πασαρέλας μεταξύ της μητρικής άδειας και άλλων μορφών γονικής άδειας. Θεωρήσαμε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι και ένας τρόπος ο οποίος θα μας επιτρέψει να βγούμε από αυτό το αδίαξοδο και εγώ θέλω να παίξω το ρόλο ενός ε, επικοδομητικού μεσολαβητή στην περίπτωση αυτή και αν η Ουγγρική Προεδρία ακόμα ή η Πολωνική Προεδρία στο μέλλον θα μπορέσουν να πείσουν τα κράτη-μέλη να ξεχάσουν το ότι έχουν ενοχληθεί από το Κοινοβούλιο και να ξεκινήσουν να ψάχνουν μια διέξοδο από αυτό το αδιέξοδο θα μπορούσαν να είναι θετικά τα πράγματα. Ξέρω ότι η Επιτροπή σας δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό της γονικής άδεια και συγκεκριμένα της άδεια των πατέρων. Η μελέτη μας για τα θέματα αυτά θα είναι έτοιμη τον... το καλοκαίρι. Θα έχουμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Υπάρχει μία ε, δυνατότητα για τη δυνατότητα άδεια για εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας έχει εξετάσει τι γίνεται στα κράτη-μέλη και κατά πόσο μπορούν να εισαχθούν αντίστοιχα μέτρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ τα πορίσματα αυτά θα είναι διαθέσιμα στο τέλος του χρόνου για την ψαλίδα αποδοχών μεταξύ γυναικών και ανδρών πιστεύω θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια καταρχήν. Γιατί δεν υπάρχει και απόλυτη συνειδητοποίηση του προβλήματος ακόμα. Όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, όλες οι προσπάθειές μας, η ημέρα παραγωγή για την ίση αμοιβή η οποία έλαβε χώρα συγχρόνως σε όλη την Ευρώπη στις 5 Μαρτίου. Όλα αυτά πρέπει να είναι πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει να ενισχύουν. Ξέρετε ότι η μέρα ίσης αμοιβή έλαβε χώρα στην, την 5η Μαρτίου γιατί αν πάρετε το μέσον όρο των αποδοχών ανδρών και γυναικών οι γυναίκες είναι σαν να ξεκινάνε να πληρώνονται μόνο στις ε, 5 Μαρτίου μέσα στο χρόνο. Είναι σαν να δουλεύουν τις προηγούμενες 63 μέρες τζάμπα, ενώ οι άντρες πληρώνονται. Επομένως, η συγκεκριμένη ημερομηνία της ημέρας ίσης αμοιβή θα εξαρτάται και από την κίνηση αυτή τη ε, διαφορά αποδοχών. Οι υπηρεσίε μου ξεκίνησαν μια μελέτη για να αξιολογήσουν τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των μέτρων που αντιμετωπίζουν την διαφορά αποδοχών ανδρών και γυναικών και αυτή η μελέτη θα δημοσιευτεί το Σεπτέμβριο του 2011 και θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο θέμα της διαφάνειας για τις αμοιβέ. Επομένως, κυρία Πρόεδρε, θα υπάρξουν όλες αυτές οι μελέτες οι οποίες θα δημοσιευθούν. Είπαμε το καλοκαίρι για την γονική άδεια των ανδρών, η, το θέμα των, διαφορών αμοιβή το Σεπτέμβριο και μετά η οδηγία για την φροντίδα εξερτημένων ατόμων στην οικογένεια το Δεκέμβριο. Ένα ακόμα σημαντικό θέμα που θέλω να αναφέρω είναι η βία κατά των γυναικών. Η δική σας ίδια <clears throat> η έκθεση κυρία Πρόεδρε θίτει πολύ σημαντικά σημεία και πιστεύω ότι και το έργο της Κομισιόν θα αντιμετωπίσει πολλές από τις ανησυχίες σας. Όπως έχουμε υποσχεθεί υπάρχει ένα πακέτο για τα δικαιώματα των θυμάτων που θα εξεταστεί το Μάιο του ενεστώτος έτους. Το πακέτο αυτό έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει ότι τα θύματα που φυσικά περιλαμβάνουν και τις γυναίκες, τα θύματα βίας, ότι θα έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους και θα έχουν την υποστήριξη και την προστασία την οποία θα πρέπει να έχουν. <clears throat> θα περιλαμβάνει το πακέτο αυτό νομοθετικά μέτρα, αλλά επίσης και μέτρα οικονομικής υποστήριξης σε ΜΚΟ, σε τοπικές αρχές, ώστε να αναπτυχθούν ε, διεθνικά σχέδια για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, των παιδιών και άλλων ατόμων. Αυτό το έργο λοιπόν είναι εν εξελίξη και πιστεύω ότι το πακέτο για τα θύματα θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και για την Επιτροπή σας. Στρέφομαι τώρα προς ένα θέμα για το οποίο έχω εργαστεί πάρα πολύ έντονα τις προηγούμενες εβδομάδες, το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στην λήψη αποφάσεων. Ξέρετε ότι εδώ είναι πάρα πολύ βραδία η πρόοδος. Έχει συζητηθεί το θέμα αυτό και στα πλαίσια της ημέρας των γυναικών. Δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και φαντάζομαι ότι έχετε δει και την δημοσίευση για την ε, ισορροπία της παρουσίας των γυναικών στις λήψεις, στη λήψη αποφάσεων και στις επιχειρήσεις. Σας είπα ε, επίσης ότι συνάντησα τους επικεφαλείς διοικητικών συμβουλίων και επιχειρήσεων οι οποίες είναι εισηγμένες στο, στα χρηματιστήρια στις αρχές του Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες για να δούμε το θέμα αυτό της συμμετοχής των γυναικών. Ο στόχος μου ήταν να τους δεσμεύσω εθελοντικά να κάνουν προσπάθειες να επιτύχουν στόχους όπως 30% το 2015 και 40% το 2020 για τη συμμετοχή γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Έχω προσκαλέσει αυτές τις εταιρείε λοιπόν μέχρι το Μάρτιο του 2012 να υπογράψουν μια υπόσχεση και μια δέσμευση προς την κατεύθυνση αυτών των στόχων και όχι μόνο να δαπανούν ωραία λόγια αλλά να έχουν και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ότι θα φέρουν τις γυναίκες σε θέσεις ηγεσία, ότι θα αντικαθιστούν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων του που απέρχονται από γυναίκες με προσόντα. Γυναίκες με προσόντα Το υπογραμμίζω αυτό. Δεν θέλουμε απλώς να έχουμε γυναίκες για την ποσόστοση. Θέλουμε γυναίκες με προσόντα που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι εκεί γιατί είναι καλές στη δουλειά τους και γιατί θα βοηθήσουν μια εταιρεία να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ενεργή στελέχωση με γυναίκες που έχουν προσόντα στο μεσαίο και υψηλό επίπεδο στελεχών είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για μας και φυσικά χαιρετίζω το σχέδιο έκθεση της κυρίας Κράτσα που αντιμετωπίζει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Και βλέπω ότι συμφωνούμε ότι, στο ότι οι μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να έχουν την πρώτη και τελευταία φυσικά ευκαιρία να κάνουν ορατά αυτά τα μέτρα υπέρ της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών και να αυξήσουν την συμμετοχή των γυναικών σε φορείς διοίκησης επιχειρήσεων μέσω μέτρων οικειοθελών. Ιδάλλως θα υποβληθούν μέτρα εκ των έξω στις επιχειρήσεις αυτές είναι ένα θέμα που αφορά τι επιχειρήσεις, αλλά όπως λέμε στα αγγλικά, women mean business. Οι γυναίκες είναι σοβαρέ για το θέμα αυτό, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και οι γυναίκες οι οποίες έχουν προσόντα υπάρχουν και βρίσκονται στην αγορά εργασία. Το θέμα είναι να τις, να τις πάρει και να τις φέρει σε μια θέση όπου μπορούν πράγματι να παίξουν κάποιο ρόλο και πιστεύω ότι οι συντονισμένε μας προσπάθειες, κυρία Πρόεδρε, θα βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε έτσι μια μεγαλύτερη πολυμορφία στις υψηλές θέσεις διοίκησης των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρέντινγκ. Είμαι πεπισμένη ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν σειρά ερωτήσεων στον τομέα που μας απασχολεί σήμερα. Θα ήθελα Ευθύς αμέσως να σας ενημερώσω ότι έχουμε προβλέψει μέχρι τις 11.30 να συνεχιστεί η συζήτηση. Δυστυχώς όμως θα χρειάζεται να αποχωρήσει στις 11 και 4 η κυρία Ρέντινγκ. Οπότε θα ήθελα και εσείς να το έχετε κατά νου για να μπορέσουμε με κοινή προσπάθεια να τηρήσουμε το χρόνο και να ακούσουμε και τις απαντήσεις ερωτήσεις που θα θέσουν οι συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ματέρα που είναι η συγγήτριά μας εδώ στην Επιτροπή για το νομοθετικό πρόγραμμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Εγώ ήθελα να κάνω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις για να πείσω και χρόνο στις συναδέλφους. Το 2008 η Επιτροπή Γυναικών ενέκρινε μία έκθεση της κυρίας Μπάουερ και ζητούσε από την Κομισιόν ειδικά μέτρα για να σταματήσει η μισθολογική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Από το 2008 μέχρι το 2011, δηλαδή σήμερα, όταν βλέπουμε να μην έχουν γίνει βήματα. Τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν για να σταματήσει αυτές τις διακρίσεις που εκθέτουν τις γυναίκες ε, στην φτώχεια. Δεύτερη ερώτηση. Διότι συζητείται το θέμα σε μερικά εθνικά κοινοβούλια μεταξύ των οποίων και το Ιταλικό, το οποίο ψηφίζει σήμερα, τις ροζ ποσοστώσεις για τη στελέχωση των επιχειρήσεων με γυναίκες. Εγώ δεν θα ήθελα βέβαια να θεωρηθούν οι γυναίκες ως κυδαιμονευόμενα άτομα τα οποία πρέπει να τα προστατεύουμε γιατί είναι ιδιαίτερα ευπαθή. Πολλές από τις γυναίκες που είναι σήμερα στο κοινοβούλιο βρίσκονται εδώ γιατί μπήκανε στην ποσόστοση των κομμάτων τους. Αλλά για να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον επιχειρηματικό κόσμο και στη δυνατότητα πρόσβασης των γυναικών Πέρα από τις γυναικείες ποσοστώσεις, κουατερόζα στα Ιταλικά, ε, έχει κάτι κατά νου η Κομισιόν για να διασφαλίσει στις γυναίκες και πρόσβαση στα πολιτικά θεσμικά όργανα. Η Γαλλία και η Ολλανδία βρίσκονται στην πρωτοπορία και η Ιταλία ελπίζω σήμερα συσπυρώνοντας όλα τα κόμματα υπέρ να κάνει και αυτή κάτι. Η Κομισιόν όμως τι θα κάνει... Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η κυρία Ματέρα το είπε πολύ ωραία ήδη προηγουμένως, γιατί ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο θέμα αυτό του χάσματος αμοιβή. Είπατε ένας βασικός λόγος είναι ότι οι γυναίκες εργάζονται με μερική απασχόληση και διακόπτουν πολλές φορές την καριέρα τους. Αλλά για τη Γερμανία βλέπουμε ότι ακόμα και αν αφαιρέσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες που έχουν να κάνουν με την μερική εργασία και με τη διακοπή της καριέρας παραμένει μια ψαλίδα, μια διαφορά 8%, 8 μεταξύ των αμοιβών ανδρών και γυναικών. Είναι μια διαρθρωτική επομένως διαφορά. Τι θα κάνουμε με αυτό το 8% που δεν έχει να κάνει με τη μερική απασχόληση και τους άλλους παράγοντες που αναφέρθηκαν. Επίσης αυτό το οποίο είπατε είναι σωστό. Πρέπει να έχουμε διαφάνεια. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις επιχειρήσεις, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για τις διαφορές σε μισθολογικό επίπεδο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μια εξτατεία και να συμπεριληφθούν και κάποιες ε, νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό που έγινε στη Βαβαρία το 2008 είναι ήδη θετικό. Μιλάτε για μελέτες, αλλά έχουν γίνει χιλιάδες μελέτες για τις διαφορές των αμοιβών. Χρειαζόμαστε ακόμα μια μελέτη για να προχωρήσουμε σε πραγματικές νομοθετικές ε, ρυθμίσεις. Έχουν υπάρξει προτάσεις εδώ και πολύ καιρό για τα θέματα αυτά. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να υπάρχει η Ευρωπαϊκή ημέρα για την ίση αμοιβή. Αυτό είναι μια ωραία όμως ε, πρωτοβουλία, αλλά στις 5 Μαρτίου δεν υπήρξε πραγματική δυνατότητα για τις γυναίκες, τις οργανώσεις τους και τα συνδικάτα να κινητοποιηθούν για τα θέματα αυτά. Και εγώ θα ήθελα όταν γίνονται εκστρατείε, τότε αυτέ οι εκστρατείε να γίνονται πραγματικά με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η Αντιπρόεδρος, η κυρία Στρέλα, θα πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην Επιτροπή μας. Για να μην χάνουμε χρόνο, θα σχολιάσω το θέμα που με απασχολεί περισσότερο, διότι είμαι εισηγήτρια για την αναθεώρηση της οδηγίας ε, σχετικά με την άδεια Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, ενέκρινε με σαφέστατη πλειοψηφία τις προτάσεις ε, που είναι επιτάπητος αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί επ' Αληθεύει επίση, όπως γνωρίζουμε, ότι το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει προσδώσει τη δέουσα σημασία στο θέμα ότι εξακολουθούν να υφίστανται πολλές δυσκολίες και πολλές ενστάσεις από πλευράς των κρατών μελών και από όσο γνωρίζω, κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας, τίποτα δεν έχει γίνει ακόμη για αυτό το θέμα. Υπήρξε μια πρώτη πρωτοβουλία Ουγγρικής ε, Προεδρίας και υπήρχαν προσδοκίες ε, ε, ότι θα έδινε μια όθηση στο θέμα η Ουγγρική Προεδρία, τόσο ώστε να περατωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Διότι οι οικογένειες, οι γυναίκες, τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν νόμιμες ε, προσδοκίες ε, για αυτό το ζήτημα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα διαβήματα που έκανε, ούτως ώστε να απεμπλακεί η κατάσταση. Πλην όμως, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει από πλευράς όλων των θεσμικών οργάνων να ε, υπάρχει μια διαλλακτική στάση, ούτως ώστε να μπορέσουμε όλοι να διαπραγματευτούμε. Στο Συμβούλιο όπως σας είπα, δεν έχει αναλυθεί καμία ε, πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας μέχρι τούδε. Ε, ελπίζουμε να δείξει καλή θέληση το Συμβούλιο και Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, Επίτροπε, δεν, μπορούμε, ε, δεν μπορούν στο Συμβούλιο να αγνοούν την πρόταση ε, του Κοινοβουλίου, διότι έχει ενισχυμένες αρμοδιότητες στο Κοινοβούλιο βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, τοποθετήθηκε, ανέλησε την κατάσταση και το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν λάβει γνώση της πρότασης του Κοινοβουλίου. Σχετικά με τη μελέτη τώρα για την άδεια πατρότητα και το δημοσιονομικό αντίκτυπο της πρότασης ε, που τώρα προωθεί η Επιτροπή και που θα είναι διαθέσιμη στην Άνοιξη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές ε, με τη μελέτη που δρομολόγησε το Κοινοβούλιο Εμείς έχουμε τα πορίσματα μιας μελέτης που ζήτησε να διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε στοιχείο για τα κράτη-μέλη και σε σχέση με την άδεια μητρότητας ή με την άδεια πατρότητας Έχουμε στοιχεία ε, σε αυτή την έκθεση. Η έκθεση δείχνει ε, ότι είχαμε μόνο αύξηση της τάξης του 1,24% μόνο της συμμετοχής των γυναικών στις ε, επιχειρήσεις ε, και είδαμε Επίσης, ότι στο, στην αγορά έργασης δεν έχουν καλυφθεί τα κενά που υπάρχουν ούτε για την άδεια μητρότητας, ούτε για την άδεια πατρότητας. Τώρα ε, υλοποιούμε την στρατηγική 2020. Ένας από τους στόχους είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να προωθηθεί εργασία στις, για τις γυναίκες. Θα κλείσω, Πρόεδρε, κάνοντας μία παρατήρηση μόνο για την θέσπιση του συστήματος των ποσοστώσεων ε, για την οικονομική δραστηριότητα και συγκεκριμένα στις διευθυντικές σχέσεις και στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Ευπρόσδεκτη η πρωτοβουλία βεβαίω. Θα ήθελα όμως να κάνω μια διάκριση αυτή. Η ποσόστος δεν αφορά στις γυναίκες αποκλειστικά, αφορά και στα δύο φύλλα έτσι συμβαίνει και στην πολιτική σκηνή. Οι κανόνε περισσότερα των φύλων ε, στο ΕΚΑ, στο τεκράτο μέλο, καλύπτουν τα δύο φύλλα. Δεν ξέρουμε ακριβώ τι θα συμβεί στο μέλλον. Μπορεί οι άντρε να χρειαστούν αυτή την ποσόστοση μελλοντικά. Ε, Κάτι άλλο τώρα. Πέρα από το ότι καλύπτει τα δύο φύλλα η ποσόστοση, αποσκοπεί στην ισότιμη εκπροσώπηση όλων και σας είπα ότι οι μελέτες δείχνουν πως ε, όπου υπάρχουν ε, γυναίκες σε ποσοστό 30% στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, ε, το κέρδος ανέρχεται σε 70% προς την κερδοφορία των επιχειρήσεων μπορούμε να πούμε ότι χρειαζόμαστε γυναίκες με προσόντα, αλλά και άντρες με προσόντα χρειαζόμαστε. Είτε μιλάμε για την κοινωνική ζωή, είτε για την επαγγελματική. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Στρέλα. Κυρία Τόμψεν τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ κυρία Ρέριν για την ε, ανακοίνωσή σας της 1ης Μαρτίου για την συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Νομίζω ότι σημαντικό το ότι αυτή η ανακοίνωση έφτασε με τις εφημερίδες στα πιο ακριτικά μέρη της Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πρώτες ύλες μας. Μιλάμε για τις πρώτες ύλες, μιλάμε για τα βασικά προϊόντα, δεν μιλάμε για τις γυναίκες. Εμείς από την Επιτροπή μας θέλουμε να αναπτύξουμε μια εκστρατεία λέγοντας ότι οι γυναίκες πραγματικά θέλουν να τις πάρουμε στα σοβαρά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουν αυτό οι επιχειρήσεις μας. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό και επίσης οι γυναίκες να έχουν πολιτική επιρροή. Έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο αλλά δεν έχουμε την αντίστοιχη οικονομική επιρροή στον οικονομικό στίβο για τη λήψη αποφάσεων και αν γυναίκε υπήρχαν στι εταιρείε χρηματοοικονομικέ, ίσω δεν θα είχαμε αντιμετωπίσει μια τόσο μεγάλη κρίση. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά το έργο τη Κομισιόν για τα θέματα λήψη απόφαση και τα δύο φύλλα. Κάτι ακόμα. Πέρσι το Μάρτιο πήρατε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με τη χάρτα για τις ε, γυναίκες που ενεκρίθη από την Κομισιόν. Κάθε φορά όμω που έχουμε μία ανακοίνωση από την Κομισιόν, είχαμε μία από τον κύριο την προηγούμενη εβδομάδα γιατί το σχέδιο αποδοτικότητα στην ενέργεια, δημιουργία πολλών θέσεων εργασία, πολύ μεγάλη απασχόληση. Δεν υπήρχε η λέξη φίλο, δεν υπήρχε η λέξη γυναίκα. Σε καμία από τι εκθέσει αυτέ που παίρνουμε από την Κομισιόν οι άλλες γενικές διευθύνσεις, οι άλλοι επίτροποι λοιπόν δεν ασχολούνται με τα θέματα αυτά, θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο για να γίνει πιο απτός αυτός ο στόχος. Θα ήθελα και εγώ ίδια να προτείνω να προσκαλέσουμε τον κύριο Ούτιγκερ εδώ, γιατί δεν άκουσε ποτέ για το φίλο και τη διάστασή του. Και επίσης το θέμα της ίσης αμοιβής. Λέμε στην οδηγία ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε για ίση απασχόληση, αλλά για εργασία ίσης αξίας. Ένα εργαλείο να το επιτύχουμε αυτό είναι η διαφάνεια. Υπάρχει όμως ένα άλλο πρόβλημα. στην χώρα μου, τη Δανία, τα συνδικάτα έχουν από κοινού διεξαγάγει μια μεγάλη μελέτη και λένε ότι υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με την ισότητα αμοιβή. Χρειάζεται η Κομισιόν να καθορίσει πότε η εργασία είναι ίση αξία. Γιατί λένε πρέπει να υπάρχει ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξια Τι είναι τώρα η εργασία ίσης αξια πω μπορούμε να μιλάμε για ίση αμοιβή χωρίς να υπάρχει ένα οδηγό για τον καθορισμό τη ίση αξία. Παραδείγματο χάρη, ένα άνδρα ο οποίο καθαρίζει έξω από το κοινοβούλιο, παίρνει πιο πολλά λεφτά από μια γυναίκα που καθαρίζει μέσα στο κοινοβούλιο. Πρέπει όμως να ξέρουμε αν αυτό το έργο είναι ίσης αξίας ή όχι. Θέλουμε λοιπόν η Κομισιόν να μας δώσει κάποια εργαλεία και κάποιους νέους ορισμούς για το τι ακριβώς σημαίνει εργασία ίσης αξίας ώστε τα συνδικάτα στην Ευρώπη να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές ως ένα εργαλείο για να επιτύχουν πραγματικά την ίση αμοιβή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. κυρία Παρανόβα τώρα. Uh, σας ευχαριστώ και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Επίτροπο για όλες τις προσπάθειες και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Γνωρίζω πολύ καλά ότι στην αρχή της εντολής σας, όταν σας θέσαμε ορισμένα ερωτήματα, είπατε ότι με μεγάλη ταχύτητα θα μας δώσετε ένα πρόγραμμα και ένα νομοθετικό πακέτο. Το ερώτημά μου είναι το εξή, σαν συνέχεια αυτό που είπε η κυρία Τόμψεν. Εάν φτάσουμε το ποσοστό των 40% των γυναικών σε υψηλές θέσεις επιχειρήσεων ή στην πολιτική, θα συμφωνούσα ότι ίσως η νομοθετική προώθηση των ποσοστών δεν θα είναι πια απαραίτητη, αλλά πόρο και παρασάγκας απέχουμε από κάτι τέτοιο. Υπάρχουν χώρες όπου η διαφορά αποδοχών ανδρών και γυναικών ξεπερνάει το 30%. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτά τα μέτρα είναι επαρκή, ότι αρκεί να λέμε σε επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν πιο πολλές γυναίκες ή χρειαζόμαστε μια πιο έντονη δράση για να υπάρξουν ποσοστώσεις και τα άλλα εργαλεία τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Και το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με τη μητρική θνησιμότητα. Αυτό φυσικά δεν απασχολεί μόνο εσάς αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια μεγάλη ανισότητα στο θέμα αυτό της μετρικής θυσιμότητας μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο μας κάνει, δυσκολεύει το να επιτύχουμε τον πέμπτο στόχο της χιλιετίας. Υπάρχει κάποια μια για το θέμα αυτό από την Κομισιόν και επίσης για το θέμα των ε, των συντάξεων και της ένδειας των γυναικών θα κάνετε κάτι για τα θέματα αυτά στη Λευκή Βίβλο. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπόσκουτ, τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Um, u heeft daar, uh, commissaris. Η Επίτροπος έκανε μια πολύ σύντομη αναφορά για τις ε, γυναίκες ε, θύματα ε, θύματα ακροτηριασμών ή εγκλημάτων τιμής και είχατε μιλήσει και για τις σχετικές ποινές. Σε αυτό το πακέτο λοιπόν προτείνεται μία στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμηθεί οποιαδήποτε μορφή βίας κατά των γυναικών και πώς σκοπεύετε να τα καταστήσετε όλα αυτά αποτελεσματικά και συγκεκριμένα. Και ρωτώ, ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον για το παρατηρητήριο κατά της βίας ε, θα συσταθεί αυτό το παρατηρητήριο για τους ακροτηριασμούς των ε, γεννητικών οργάνων ε, των ε, γυναικών. Εσείς είχατε εξαγγείλει μια στρατηγική για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Τι κάνατε σχετικά. Επίσης, για το Ιστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων θα διαμορφώσει συγκεκριμένους δείκτες για να μπορέσουμε να μελετήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Μποσκούτ. Η κυρία Μπίσκεβιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την πρωτοβουλία σας ε, σχετικά με την ε, αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Θα ήθελα όμως να σας θέσω μια ερώτηση για την θέση που κατέχουν οι γυναίκες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν θεωρείτε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αναλάβει μία πρωτοβουλία σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων για τις διευθυντικές θέσεις των γυναικών στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα δώσουμε και το παράδειγμα εφόσον τώρα πραγματευόμαστε το θέμα της εκπροσώπησης των γυναικών στις επιχειρήσεις και ζητούμε αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξή Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαγγείλει ένα το καταπολέμησης της ε, βίας ε, κατά των γυναικών. Ε, το Κοινοβούλιο το έχει ζητήσει επανειλημμένα. Και τρίτη ερώτηση. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η οδηγία για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης έχει παραγωνιστεί η οδηγία, κατά τη γνώμη μου, διότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντική η οδηγία για την ισότητα των δύο φύλων. Πιστεύετε ότι θα ε, καταλήξουμε κάπου με αυτήν την οδηγία. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Σοβή. Αξιότιμη Πίτρουπ, σας ευχαριστώ για τις εργασίες ε, των τελευταίων ετών. Σας έχω ακούσει ε, ε, επανειλημμένα με μεγάλο ενδιαφέρον και ξέρω πόσο αφοσιωμένοι είστε στη δουλειά σας σχετικά με την ισότητα των δύο φίλων. Εδώ και δεκαετίες συζητούμε και εξετάζουμε αυτό το θέμα. Θα θέσω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα επ' αυτού. Στο άρθρο 2 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται η προστασία της ισότητας των δύο φύλων και στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων επίσης υπάρχει μια παρεμφερή σε διάταξη προπενταετίας κατά τη διάρκεια ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, υπήρξε και επίσημη υποστήριξη από τους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων για αυτήν την ιδέα. Ε, ξέρουμε όμως ότι δεν δόθη συνέχεια γιατί στο μεταξύ δεν είναι τα ίδια άτομα που κατέχουν αυτά τα υψηλά αξιώματα. Θα ήθελα να ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την τροποποίηση της κείμενης ε, νομοθεσίας. Ε, χρειαζόμαστε αποτίμηση της κατάστασης και συγκεκριμένα μέτρα ώστε οι κείμενες διατάξεις να υλοποιηθούν, να εφαρμοστούν σωστά. Ε, ποιες συστάσεις ε, θα είχατε να εισηγηθείτε για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε κύριε Οβέρ, Πρόεδρος. Ε, τώρα η κυρία Ρονέρο Λόπερς τώρα. τώρα Gracias, Presidenta. Gracias, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Ρέντινγκ. Θέλω να σταθώ και εγώ στο θέμα της κυρίας Μποσκούτ για τη βία κατά των γυναικών, διότι ο Ούγγρος Υπουργός Δικαιοσύνης όταν τον ρώτησα για τη βία κατά των γυναικών, ε, για τον αριθμό των ε, δολοφονημένων γυναικών στην Ουγγαρία, δεν είχε τον αριθμό. Αυτό στην Ισπανία θα ήταν ανήκουστο, διότι υπάρχει... Αυτό βγαίνει σε εφημερίδες, ε, διότι γίνεται, μεσολαβεί πάντα μια τεράστια κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και είναι κρίμα που υπάρχουν χώρες που δεν έχουν ευαισθησία στις, ε, ε, κατά της βίας για τις, των γυναικών. Τι κάνει το παρατηρητήριο ε, για την ε, βία κατά των γυναικών. Η διευθύντρια του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων δεν είχε πληροφορίες για αυτό το θέμα. Τι θα γίνει με αυτό το παρατηρητήριο λοιπόν. Θα λειτουργήσει, πού θα λειτουργήσει. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε τα στοιχεία και αυτό γιατί δεν έχουμε το παρατηρητήριο. Ξέρετε ότι εγώ με την ε, κυρία Χιμένες ε, συμμεριστήκαμε την έκθεση για τις ε, γυναίκες, για, την, για τις επιπτώσεις ενός ε, μηχανισμού για την ε, προστασία ε, των γυναικών. Λοιπόν, ποιες επιπτώσεις έχουμε εδώ, ετοιμάζουμε αυτό το πακέτο για τα θύματα, μια έκθεση για τα θύματα. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε πόσοι νόμοι προστασίας ισχύουν σήμερα στην Ευρώπη και τι θα συμβεί με το πακέτο που μας αναγγείλατε ότι θα ήταν έτοιμο την άνοιξη και καθυστερεί. Γιατί καθυστερεί αυτό το πακέτο για τα θύματα. Και πότε τελικά θα μας έρθει εδώ στο Κοινοβούλιο. Και τι θα συμβεί με τις χώρες εκείνες ε, που έχουν είτε αστική διαδικασία είτε ποινική διαδικασία και δεν έχουν μεικτή διαδικασία, πώς ε, θα υπάρξει αναγνώριση της αστικής ευθύνης. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι έχουμε ακόμη 11 συναδέλφους στον κατάλογο. Σας παρακαλώ, σας θέρμο παρακαλώ να αυτοπεριοριστείτε να μην υπερπαίνετε το χρόνο στις ε, παρεμβάσεις σας. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Γιαβελέσκα και κατόπιν θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο Ρέντινγκ για να απαντήσει στο πρώτο γύρο ερωτήσεων. Παρακαλώ το τονίζω, ε, έχουμε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, παρακαλείστε να το έχετε και εσείς κατά νου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο τον πιο σύντομη. Πιστεύω ότι η Πολωνία όταν αναλάβει την Προεδρία θα μπορέσει το ταχύτερο δυνατό να καταλήξει σε μια συμβαστική λύση για την πατρική άδεια. Στην έκθεση αυτή επίσης μιλήσαμε για την άδεια υιοθεσία. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Είναι πολύ καλό να δώσουμε έμφαση στο θέμα τη άδεια για τι γυναίκε. Σκεφτείτε και τι μητέρε που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και υποχρεώνονται να υιοθετήσουν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια σχέδια για το θέμα αυτό ή κάποια λύση ή κάποιες ελάχιστες λύσεις για την άδεια υιοθεσία. Γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές για τα θέματα αυτά. Στην Πολωνία το 2007 μια γυναίκα που υιοθετεί ένα παιδί πάνω από 12 μηνών ηλικίας δεν μπορεί να πάρει ούτε μια μέρα άδεια υιοθεσία. Ενώ στην Πολωνία τώρα έχουμε, ε, έχουμε πολύ μεγαλύτερη άδεια μητρική και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιες προτάσεις για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο Ρέντινγκ τώρα για να απαντήσει σε αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ε, παρακαλώ. Πρόεδρε, Επιτρέψτε μου να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις, διότι ε, κάποια μέλη της Επιτροπής σας ε, έθεσαν ερωτήσεις ίδιου τύπου. Ας ε, ξεκινήσω με το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Υποσχέθηκα ένα πακέτο για τα θύματα την Άνοιξη. Εξ αρχής είχα υποσχεθεί αυτό το εαρινό πακέτο και θα έρθει την Άνοιξη αυτό το πακέτο όντως. Στις 11 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά. Θα εμπεριέχει νομικά μέτρα και οικονομικά μέτρα. Επίσης θα εμπεριέχει έναν οδικό χάρτη. Το τέστην δεν θα είναι μια άπαξ δράση, θα προγραμματίσουμε για το μέλλον όλες τις εργασίες μας στον τομέα αυτό. Ένα συγκεκριμένο ερώτημα τώρα για το ένταλμα, την εντολή προστασίας. Θα υποβάλω νομοθετική πρόταση για μέτρα αστικού δικαίου. Έχετε ε, αναχείρασε μια πρόταση για τα μέτρα ποινικού δικαίου. Αν υπάρξουν τροποποιήσεις για την υφιστάμενη πρόταση, τότε θα έχουμε δύο σχέδια. Το παλιό κείμενο για το ποινικό δίκαιο, το νέο για το αστικό και τα δύο μαζί θα καλύπτουν πλέον όλες, όλα τα νομοθετικά ενδεχόμενα που πρέπει να καλύψουμε ούτως ώστε ε, να κατοχυρώσουμε μια ουσιαστική, μια πραγματική προστασία ακολουθούν ε, οι προτάσεις στη σωστή κατεύθυνση. Συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο και οι τροποποιήσεις ε, του σχεδίου, Πρόεδρε, είναι λιγοστές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προχωρήσει ταχύτατα η διαδικασία. Υπάρχει και άλλη εναλλακτική λύση βεβαίως. Να καταθέσω πρόταση και για τα, τις αξιόπινες πράξεις, για εγκλήματα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι απαραίτητο, διότι ε, μπορεί να αρκέσουν κάποιες ε, τροπολογίες που ήδη έχουν κατατεθεί για τα προηγούμενα σχέδια. Αναμένονται συγκεκριμένε δράσεις. Κατόπιν, τώρα γενετικών γεννητικών οργάνων, ε, γυναικεία περιτομή. Το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Δύο Φύλων καλείται να μας παρουσιάσει τα στατιστικά δεδομένα, να προβεί στην ανάλυση του ζητήματος ε, και το θέμα αυτό καλύπτεται στον οδικό χάρτη για τα δικαιώματα των θυμάτων. Όταν έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα ε, στοιχεία ε, όταν τα λάβουμε δηλαδή από το Ινστιτούτο για την ισότητα των δύο φύλων, θα προχωρήσουμε κατά πάσα πιθανότητα το 2012, υποβάλλοντας πλέον την νομική, την νομοθετική πρόταση. Α, το 2013 διορθώνει η ομιλήτρια για την νομική πράξη. Θα περιμένουμε το 2013 χρειαζόμαστε την ανάλυση από το Ινστιτούτο Ισότητας των δύο φύλων. Επίσης ζήτησα από αυτό το Ινστιτούτο να μας ε, προσκομίσει τα δεδομένα για την βία κατά των γυναικών και το Ινστιτούτο της Ευγέννηση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Ισότητας των Δύο Φύλων για αυτό το θέμα. Εγώ μετέβην και στα δύο Ινστιτούτα και επέμεινα να φροντίσουν ώστε να μην υπάρξει επικάλυψη εργασιών. Επικουρούν το ένα το άλλο για αυτά τα δύο ζητήματα, ακροτηριασμός των γυναικείων γενετικών οργάνων και βία κατά των γυναικών. Αυτά τα δύο σημεία είναι σημεία προτεραιότητας και για τα δύο Ινστιτούτα και θα επιτελέσουν το έργο τους. Το θέμα τώρα της μισθολογικής διαφοράς ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Το μισθολογικό κενό, χάσμα. Ε, ξεκίνησα τις εργασίες ε, για την διαφάνεια, διότι με τις εκστρατείες διαφάνειας ε, και ενημέρωσης μπορούμε να προχωρήσουμε και να περιστήλουμε το, τη μισθολογική διαφορά. Αυτή τη στιγμή εξετάζω αποτελέσματα, αναλύω μάλλον τα αποτελέσματα των προηγουμένων εκστρατιών. Το 2009, το 2010 είχαμε μια αντίστοιχη εκστρατεία και συνεργαστήκαμε με Ινστιτούτα, συνδιοργανώσαμε τις εκστρατείες με τα Ινστιτούτα. Έχουμε 308 οργανώσεις εταίρους σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεργάζονται μαζί μας και ε, διάκυνται μάλλον θετικά ως προς ε, την αποτελεσματικότητα τέτοιων εκστρατιών ενημέρωσης ήλθα σε επαφή μαζί τους ε, για να προετοιμάσω την ε, Διεθνή ημέρα του 2012 για την ίση αμοιβή. Φέτος δοκιμάσαμε για πρώτη φορά αυτό το σύστημα, δηλαδή και προετοιμαζόμαστε ήδη από τώρα για το 2012 σε συνεργασία με αυτές τις οργανώσεις εταίρου. Ε, μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα δεν ικανοποιηθήκατε από το 2011 ούτε και εγώ, αλλά θα προετοιμαστούμε καλύτερα για το 2012. Έχουμε άπλετο χρόνο μπροστά μας για να προετοιμαστούμε, να, έχουμε, να δράσουμε με πυγμή του χρόνου. Είναι μια καλή ιδέα, οι άνθρωποι μας ακούν, οι οργανώσεις ε, ε, εταίροι θα μας συνδράμουν και θα ε, φέρουν αυτή την πυγμή που χρειαζόμαστε και ταυτόχρονα θα έχουμε και ενημερωτικό υλικό για τις εκστρατείες και σύντομα θα είναι διαθέσιμο το υλικό μάλιστα, μπορείτε να το δείτε. Ας περάσω τώρα στην αδία μητρότητος τα πράγματα έχουν ε, όπως έχουν, το γνωρίζετε. Ε, εσείς υπερψηφίσατε μία έκθεση, γνωρίζετε ακριβώ το περιεχόμενο της έκθεσης και το Συμβούλιο αρνείται. Αυτή είναι η κατάσταση αν όλοι μένουν οχυρωμένοι και μένουν στη θέση τους, δεν θα σημειωθεί η πρόοδος. Η Βελγική Προεδρία ήδη προσπάθησε να έρθει σε επαφή με κάποια από τα κράτη-μέλη, αλλά αρνήθηκαν. Η Ουγγρική Προεδρία επίσης διοργάνωσε ε, συνεδριάσεις, συναντήσεις για να γίνουν όλα πιο ομαλά. Τίποτα, αμετακίνητα είναι τα κράτη-μέλη στη θέση τους ε, προς το παρόν. Εγώ τι μπορώ να προσπαθήσω να προσεγγίσω ε, με διαφορετικό τρόπο το θέμα. Αν ε, το Συμβούλιο εξετάζει την έκθεση του Κοινοβουλίου, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Οπότε σκεφτήκαμε μία άλλη διέξοδο, ούτω ώστε να μετακινηθούν οι μεν και η δε από τις θέσεις τους. Η Πολωνική Προεδρία που προωθεί το όλο θέμα της μητρότητας το είχε αναδείξει σε ε, ε, μεγάλη προτεραιότητα μπορεί να αναλάβει μια δράση που θα τελεσφορήσει. Θα ήθελα μόνο να σας ζητήσω να μην, ε, να μην δείχνετε πείσμα για τη δική σας τη θέση. Όλοι θα πρέπει να, να ε, φανούν πιο διαλλακτικοί, ακόμη και το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό το λόγο σας είπα Ας ξεκινήσουμε ε, τη συζήτηση για τη ρήτρα, την επωνομαζόμενη πάσερελη, δηλαδή τη μεταβατική ρήτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ρήτρα, διότι θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη, τα πιο αδιάλακτα κράτη-μέλη, θα τα βοηθήσει να αρχίσουν τη συζήτηση, να αρχίσουν το διάλογο. Ας προχωρήσουμε με αυτήν τη ρήτρα και να διαπιστώσουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Η μόνη διέξοδος, ε, κατά αυτή είναι. Ε, προφανώς θα επανέλθουμε και θα σας ενημερώσουμε για τις μελλοντικές εξελίξεις. Ως προς τις ποσοστώσεις δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες ε, διότι εκτενέστατα σας έχω σχολιάσει ε, τα περί ποσοστώσεων. Ο στόχος είναι σαφής, η ημερομηνία είναι σαφής. 8 Μαΐου 2012 είναι η καταληκτική ημερομηνία στο ενδιάμεσο διάστημα επεξεργάζομαι ε, τα νομοθετικά, τα νομοπαρασκευαστικά σχέδια για να είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί το 2012. Από σήμερα όμως μέχρι το 2012 θα προσπαθήσω να ε, κάνω τις μεγάλες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες να εκδηλωθούν δημοσίως. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες στον οικονομικό τύπο βλέπω διαρκώς το εξής. Καθημερινά μεγάλες εταιρείες ε, εξαγγείλουν ότι μία γυναίκα ανέλαβε ένα ανώτατο αξίωμα. Αλλά δεν επαρκούν αυτές οι κινήσεις. Είναι, ε, υπάρχει κάποια δράση αλλά όχι συστηματική. Μόνο σκόρπια αποτελέσματα έχουμε προς το παρόν θα θέλαμε ένα μαζικό κίνημα. Αν εκδηλωθούν πολλέ πολλές τέτοιες συγμένε εταιρείε, θα έχουμε θετική πρόοδο τους επόμενους μήνες. Οφείλουμε εμείς να τροφοδοτούμε αυτό το κίνημα για να μην σταματήσει. Ε, πραγματικά παίρνουμε στα σοβαρά αυτό το θέμα. Είναι επίσης σημαντικό να πω το εξή. Λοιπόν, μιλάμε για το ρόλο των γυναικών στην πολιτική. Πολύ ωραία. Εγώ με την ιδιότητα της Επιτρόπου δεν μπορώ να πραγματευτώ αυτό το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική. Αυτό είναι θέμα πολιτικής ομάδας. Άλλο τι κάνω εγώ στο πολιτικό μου κόμμα, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την ιδιότητα της Επιτρόπου για να ε, προωθήσω αυτό το θέμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι σε εσωτερικό επίπεδο να κινηθώ και αυτό κάνουμε. Ε, συνειδητά έχουμε κάνει κάποια βήματα, δηλαδή οι γυναίκες στις ε, διευθυντικές θέσεις των επιχειρήσεων, 95... 4%. 22% το 2009. Από τα 4 στα 22 είναι μια μεγάλη αλλαγή. Σε 15 χρόνια. Για τα μεσαία στελέχη έχουμε διπλασιάσει το ποσοστό των γυναικών Μέχρι το 2014, αν θέλει ο Θεός, η Κομισιόν θα έχει 25% ανώτατες διοικητικές θέσεις που καλύπτονται από γυναίκες. Αυτός είναι ο στόχος μας και προχωρούμε προς τα εκεί μέρα και νύχτα. Αυτό σημαίνει 30% από, τις, από τους διορισμούς για να αντικαταστήσουμε τους αποσυρώμενους και αφιπηρετούντες θα πρέπει να είναι γυναίκες. Εάν το κάνετε αυτό νοιαστά, με έναν τρόπο που είναι συνειδητός, τότε αντιμετωπίζετε ένα διαφορετικό πρόβλημα το οποίο έχω εγώ τώρα στη γενική μου διεύθυνση. Και ξέρω ότι πρέπει να προχωρήσω στη στελέχωση τη δική μου γενική διεύθυνση, Έχω 80% γυναίκε σε ανώτερε θέσει και 70% γυναικών <clears throat> στα μεσαία στελέχη που σημαίνει πρέπει να εφαρμόσω ποσοστώσει υπέρ των ανδρών γιατί δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί. Τι δείχνει όμως αυτό. Δείχνει ότι, ότι μπορούμε να βρούμε τις γυναίκες. Αν τις ψάξετε θα τις βρείτε. Το άρθρο 18, η οδηγία του άρθρου 18 είναι σε αδίέξοδο αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω καμία δυνατότητα να βγούμε από αυτό το αδίέξοδο. Γιατί εφαρμόζεται εδώ ο κανόνας της ομοφωνίας και κάποιες από τις μεγάλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Κάθε φορά που βλέπω τους αρμόδιους υπουργούς μιλάμε για το θέμα αυτό και δυστυχώς μου λένε νιέτ, δεν γίνεται τίποτα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να βρούμε κάποια διέξοδο. Εγώ σκέφτομαι να αντιμετωπίσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα αυτής της ε, οδηγίας για, τους, ε, για τα άτομα με αναπηρίες και να παρουσιάσουμε κάποιο νομοθέτημα προς την κατεύθυνση αυτή. Εδώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια κίνηση, να προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλά το άρθρο 19 ως έχει δεν θα υπάρξει εκεί καμία πρόοδος. Δυστυχώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σινκλέρα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία μεταξύ μας στο ότι θέλουμε να σταματήσει να υπάρχει αυτή η ψαλίδα αποδοχών. Όλοι πιστεύουμε στην ισότητα των φίλων. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε μία νομοθεσία για την ίση αμοιβή το 1970, το πρώτο βιομηχανικό έθνος το οποίο έπραξε ούτως και αυτό φυσικά πρωτού μπει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά 41 χρόνια αργότερα εξακολουθούμε να έχουμε ανισότητα στην πραγματικότητα. Αυτό δείχνει ότι δεν γίνεται μόνο με νομοθεσία να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις κοινωνικές συνθήκες. Υπήρξε μια απόφαση πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ασφάλειες αυτοκινήτων. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα υπερβολικής νομοθεσίας που παράγει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Όπως λέγαμε χθε, οι ασφαλιστικές εταιρείε δεν θα μειώσουν τα ασφάλιστρα των ανδρών στο επίπεδο των γυναικών, θα αυξήσουν τα ασφάλιστρα των γυναικών στο επίπεδο των ανδρών. Επομένως, σε μια εποχή λιτότητος και περιστολής δαπανών, ουσιαστικά μια τέτοια απόφαση κοστίζει τις γυναίκες περισσότερο. Έχετε ένα αντιπαραγωγικό μέτρο το οποίο προκύπτει από την προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα της ισότητας. Για τις ποσοστώσεις και τα λοιπά, θέλω να θέσω το ερώτημα. Η Κομισιόν πιστεύει ότι πρέπει να νομοθετούμε για να οδηγήσουμε σε κάποια θύματα. Είναι θετική διάκριση η επιβολή ποσοστώσεων που οδηγεί σε κάποια θύματα. Εμείς πρέπει να είμαστε εναντίον των διακρίσεων. Αλλιώς προξενείτε θύματα. Δημιουργείτε μόνοι σας διακρίσεις. Και νομίζω θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας ε, πληροφορήσω ότι στις 11 και 10 πρέπει να ολοκληρώνουμε διότι η Αντιπρόεδρος θα πρέπει να φύγει και διάφοροι μου έχουν ζητήσει ήδη το λόγο. Μα και εγώ ήδη εξάλλου ζήτησα το λόγο, αλλά δεν θα τον πάρω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η κυρία Φιγκερέιδο έχει τώρα το λόγο και ακόμη μία τοποθέτηση. Εγώ βέβαια θα καλέσω και πάλι την Επίτροπο να έρθει στην Επιτροπή μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μια άλλη φορά για να μπορέσει η Επίτροπος να φύγει στην ώρα της. Η κυρία Μπάουερ και μετά η κυρία Φιγερέιδο. Σας ευχαριστώ λέει, κυρία Μπάουερ, δύο σύντομες ερωτήσεις και μόνο. καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την παρουσία σας σήμερα, τη χαρά μου. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μπορούμε επί εθελοντικής βάσης και μόνο να επιτύχουμε κάποια διαφάνεια. Λαμβάνοντας υπόψη την αναποτελεσματική νομοθεσία του τελευταίου αιώνα. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι αν αντιμετωπίζετε το θέμα των φορέων ισότητος. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των θέσεων των διαφορετικών φορέων ισότητας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και κλείνω. Δεν δε, δε, δε λέω τίποτα περισσότερο γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκερέντου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και σας κυρία Επίτροπε για τα ερωτήματα τα οποία τέθησαν εδώ. Απλώς ένα σύντομο σχόλιο. Για την μητρική και πατρική άδεια, το σχέδιο αυτό το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε κύριε Επίτροπε ότι έχετε εδώ την υποστήριξη της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου για να επιμείνουμε σε αυτή τη θέση του Κοινοβουλίου η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης προς το Συμβούλιο. Από την άποψη αυτή είναι σαφές ότι τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν από αυτή την πίεση μπορούμε να δούμε πέραν αυτών τι άλλες ενέργειες μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε και μεγαλύτερη υποστήριξη και μεγαλύτερη ορατότητα στο πρόβλημα αυτό. Ακριβώς πιέζοντας τα κράτη-μέλη τα οποία προσπαθούν να μποϊκοτάρουν την πρόοδο αυτής της διαδικασίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι βραχυπρόθεσμα η παρουσία σας εδώ μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να μας δώσετε μια απάντηση, να μας δώσετε την απάντηση που πήρατε από το Συμβούλιο και να κάνετε ένα απολογισμό των θέσεων του Συμβουλίου. <clears throat> Δεύτερον, για το θέμα των διακρίσεων στο χώρο εργασίας, που δεν είναι μονάχα μισθολογικού χαρακτήρα και δεν είναι μονάχα άμεσες διακρίσεις. Η κυρία Τόμσεν ήδη αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα το οποίο και εγώ έχω θίξει πολλές φορές, που είναι το θέμα της πραγματικής αξίας που θα πρέπει να έχει το έργο της γυναίκας. Τα επαγγέλματα, τα γυναικεία και οι δραστηριότητες των γυναικών θεωρούνται υποβαθμισμένες. Είναι επίγον να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες που υπάρχουν ήδη. Έχουμε ήδη παρουσιάσει προτάσεις για την αναβάθμιση της εργασίας των γυναικών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βασιστεί σε αυτές τις μεθοδολογίες και με στεναρό τρόπο να προχωρήσει σε μέτρα για τα θέματα αυτά και επίσης και οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συμβούλους ισότητος <clears throat> ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια σε πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που είχαν λάβει, με, ε, χώρα στα πλαίσια της πρωτοβουλία Equal. <clears throat> Ξέρετε ότι υπάρχει το Ίδρυμα αυτό για την ισότητα το οποίο έχει δημιουργηθεί, αλλά και μαζί με αυτό το Ίδρυμα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε σε λειτουργία μια σειρά από πρωτοβουλίες για τα θέματα αυτά. Ξέρετε επίσης ότι η διάκριση κατά των γυναικών και η ένδυά τους οφείλεται και στην επισφαλή εργασία η οποία πολλαπλασιάζει τα προβλήματα και εδώ θα ήθελα να μου απαντήσετε κυρία Επίτροπε. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Ρέντιν για να απαντήσει για τα θέματα αυτά και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να δώσω λόγο σε, το λόγο σε όλες σας. Ίσως κάποια άλλη στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε μια συζήτηση με την κυρία Ρέντιν. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω στο βαθμό του δυνατού να δώσω κάποιες απαντήσεις στο θέμα παραγωγής αυτό που αναφέρθηκε για τις ασφάλειες των αυτοκινήτων. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δείχνει τη σημασία της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όταν νομοθετούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι λέει τώρα αυτή η απόφαση του δικαστηρίου. λέει ότι το να συνδέονται τα ασφάλιστρα μόνο με το φύλλο του ασφαλιζόμενου, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Αυτό σημαίνει πραγματικά για τις ασφάλειες αυτοκινήτων, αν οι άνδρες πληρώνουν περισσότερο επειδή μόνο είναι άνδρες και για τις ασφάλειες ζωής όπου οι γυναίκες πληρώνουν περισσότερο επειδή είναι γυναίκες, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Πρέπει να εκτιμήσετε τον ατομικό κίνδυνο που επέχει ένας ασφαλιζόμενος και όχι μονάχα τα ασφάλιστρα να συνδέονται με το φύλλο στο οποίο ανήκει ο ασφαλιζόμενος. Θέματα όπως είναι το βάρος, η ηλικία, η προσωπική ιστορία, το ιστορικό ασθένειας. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη και όχι μονάχα μια συλλήβδη αντιμετώπιση επί τη βάση του φύλου. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν καιρό μέχρι το τέλος του 2012 για να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο νομικό πλαίσιο. Εγώ θα έρθω σε επαφή με τους επικεφαλείς των ε, ασφαλιστικών εταιριών το Σεπτέμβριο εφέτος για να μπορέσουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί διαφάνεια και αναλογικότητα για την εφαρμογή αυτών των μέτρων ώστε να έχουμε μια ισορροπημένη αντιμετώπιση. Για τις ποσοστώσεις τώρα. Το είπα και το ξαναείπα. Δεν είναι πανάκια οι ποσοστώσεις, δεν είναι αυτός σκοπός, μπορούν να είναι όμως ένα εργαλείο, αν δεν βλέπουμε άλλο τρόπο να εξασφαλίσουμε κάποια πρόοδο. Και εδώ φυσικά η αρχή της αναλογικότητας παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι μια απέτηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και για οποιαδήποτε πράξη θετικού χαρακτήρα η οποία πρέπει να είναι ισοδίκαια. Πρέπει να λάβουμε φυσικά υπόψη και τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα θέματα ισότητα ανδρών και γυναικών. Επί τη βάση αυτή εργάζομαι μαζί με του νομικού μα συμβούλου για να μπορέσουμε να έχουμε την βέλτιστη και στεναρότερη νομική βάση η οποία θα είναι και η βάση της επιβολής ποσοστώσεων, εάν χρειαστεί να πάμε προς την κατεύθυνση αυτή. Για την πατρική άδεια Ξέρετε ότι η Κομισιόν δεν θέλει η πατρική άδεια αυτή να τεθεί στην οδηγία για τις έγκυες εργαζόμενες. Είναι περισσότερο συνδεόμενη με τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας. Παρόλα αυτά αποφασίσαμε να εξετάσουμε τα υπέρ και τα κατά, το κόστος και το όφελος οποιασδήποτε διάταξης για την πατρική άδεια. Επομένως, να είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί να λάβουμε νομοθετικές ρυθμίσεις. Ξέρετε ότι η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να κάνει μια σημαντική αξιολόγηση αντικτύπου πριν από οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση που κάνει για, τα, για, την για τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο αυτής της νομοθεσίας. Αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως προτού η Κομισιόν λάβει κάποια απόφαση για τα θέματα αυτά. Για το πώς θα προχωρήσουμε τώρα για τη μητρική άδεια χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό ή τσατσά. Και ο παρτενέρ σας εδώ δεν είναι η Κομισιόν, είναι το Συμβούλιο. Προσπαθήστε λοιπόν να χορέψετε τάγκο. Σας ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε Ρέντινγκ. Ήθελα μόνο να διαπιστώσω ότι ε, σε σχέση με την αρχική ημερήσια διατήρηση είχαμε προβλέψει μια μισή ώρα για αυτή τη συζήτηση, αλλά αναγκαστήκαμε να τροποποιήσουμε το σχέδιό μας. Ε, περιορίσαμε το χρόνο σε μία ώρα και 15 λεπτά. Ζητώ συγγνώμη από τους αδέλφους που δεν θα έχουν χρόνο να θέσουν ερωτήματα. Ταυτόχρονα διαπιστώνω ότι όντω δεν επαρκεί μία ώρα και ένα τέταρτο για να συζητήσουμε τόσο σημαντικά ζητήματα με την Επίτροπο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μεταγενέστερα να βρούμε μια άλλη ευκαιρία για να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Πάντως ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση. Και τώρα έχουμε άλλο ένα θέμα μόνο στην ημερήσια διάταξή μας είναι η έκθεση της κυρίας Κράτσα Τσαγκαροπούλου. Οι γυναίκες και η ηγεσία επιχειρήσεων είναι ο τίτλος της έκθεσης. Και αυτή η έκθεση ε, σχετίζεται άρρηκτα με το θέμα ε, του διαλόγου μας με την κυρία Ρέντινγκ σήμερα. Και θέλουμε να συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση και θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Κράτσα να αρχίσει τη συζήτηση παρουσιάζοντας το σχέδιο έκθεσής της. Παρακαλώ κυρία Κράτσα. κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, η έκθεση στο, το σχέδιο έκθεση το οποίο συζητούμε τώρα είναι πολύ συνδεδεμένο, άμεσα συνδεδεμένο με, το, με τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως με την ε, Αντιπρόεδρο την κυρία Ρέντινγκ. Ε, είναι δηλαδή πώς θα αυξήσουμε, θα συμβάλλουμε ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις στο, ο, στις επιχειρήσεις. Ε, προσπάθησα στην έκθεση να αναδείξω την ε, πρόκληση που αποτελεί αυτό το θέμα για μια καλύτερη κοινωνία με μεγαλύτερη δικαιοσύνη και σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών ε, και παράλληλα με τη σημασία που έχει η πρόκληση αυτή για την ευρωπαϊκή οικονομία κυρίως την, την εποχή αυτή που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Έτσι λοιπόν, ε, ε, στην έκθεση, ε, η έκθεση κάνει μια παρουσίαση των, της κατάστασης των γυναικών στο, στις διευθυντικές θέσεις, πώς έχει σήμερα στην Ευρώπη ε, ε, παρουσιάζεται το χαμηλό ποσοστό των γυναικών που είναι σε θέσεις ε, προέδρων γενικών διευθυντών. Παρουσιάζεται όμως και παράλληλα οι προσπάθειες που έχουν γίνει προς την ανατροπή αυτής της κατάστασης, προσπάθειες οι οποίες έχουν να κάνουν με πρωτοβουλίες ή των επιχειρήσεων ή δικτύων γυναικών στελεχών στις επιχειρήσεις. Βλέπουμε λοιπόν πραγματικά ότι υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση, υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση, υπάρχουν προγράμματα ε, ε, ε, συμπαράσταση στην ανέλυξη των γυναικών μέσα στις επιχειρήσεις. Υπάρχει η δραστηριοποίηση των ίδιων των γυναικών με ανταλλαγή καλών πρακτικών, με ε, συνεργασία με συναδέλφους τους από τις διάφορες επιχειρήσεις, να αναδειχθεί αυτή η πρόκληση και βλέπουμε ότι έχουν, υπάρχουν και δειλά βήματα α, θετικά. Παρόλο όμως αυτή την κινητοποίηση δεν υπάρχει κάτι, ε, κάτι ενθαρρυντικό που μας πείθει ότι πρέπει να συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, ενθαρρυντικά βήματα έγιναν όταν χώρες απεφάσισαν ότι θα πάρουν πολιτικές πρωτοβουλίες και δι πρωτοβουλίες νομοθετικές δεσμευτικές. Ακόμη και προτού εφαρμοστεί ο νόμος, βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται προς αυτή τη νέα κατάσταση που τίνει να δημιουργηθεί, δηλαδή της υποχρεωτικής συμμετοχής ποσοστού γυναικών στις επιχειρήσεις και παίρνουν πρωτοβουλίες. Το πρώτο τέτοιο παράδειγμα που έχουμε στον ευρωπαϊκό χώρο, έστω και εκτός Ένωσης, είναι η Νορβηγία, η οποία έχει ένα νόμο από το 2004 σε εφαρμογή, με σαφή αποτελέσματα αυτής της, ε, με αποτελέσματα της ε, αύξησης ε, Τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα που λαμβάνονται αποφάσει. Παράλληλα όμως έχουμε και στον χώρο της Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοβουλίες, έχουμε τον νόμο στην Ισπανία, έχουμε τον νόμο πρόσφατα που ψηφίστηκε στην Γαλλία, Έχουμε την ε, συζήτηση η οποία είναι σε όριμο στάδιο στην Ιταλία. Επίσης στη Γερμανία, σε μια χώρα που υπήρχε ε, μια άρνηση ε, στην ε, εισαγωγή ποσοστώσεων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συζήτηση και σε επίπεδο μοσπονδιακής κυβέρνησης και σε επίπεδο κρατηδίων, παραδείγματο χάρη από την, υπουργό, την αρμόδια υπουργό στο, στην Μπαβιέρα. λοιπόν, όλα αυτά τα δήματα, όλα αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια ευρύτερη συνειδητοποίηση ε, της ανάγκης ενός γεγονότος μιας κατάστασης που θα δώσει μια ουσιαστική όθηση στη συμμετοχή των γυναικών και μια πραγματική δέσμευση από την πλευρά των επιχειρήσεων. Η προβληματική μας λοιπόν που αναδεικνύεται από, αυτό το, από αυτή την έκθεση είναι πώς αυτή τη δυναμική που ήδη υπάρχει και ε, τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε κράτη-μέλη θα τις αναδείξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί? Διότι υπάρχουν κάποιες περιοχές, στις οποίες, ενώ κάποιες χώρες, στις οποίες δεν γίνεται συζήτηση. Δεν γίνεται συζήτηση ούτε σε πολιτικό επίπεδο, ούτε υπάρχουν νομοθετικέ πρωτοβουλίε, ούτε οι επιχειρήσει έχουν μια τέτοια κουλτούρα που από μόνε του παίρνουν πρωτοβουλίε. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η δυναμική και αυτέ οι εμπειρίες θετικέ που έχουμε σε, από τη μια μεριά σε επίπεδο, ε, επαναλαμβάνω, ε, πολιτικών πρωτοβουλειών και νομοθετικών και από την άλλη σε επίπεδο καλών πρακτικών κάποιων επιχειρήσεων να τους δώσουμε μια προστιθεμένη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η, Το... η στιγμή που γίνεται αυτή η συζήτηση είναι ε, πολύ, ε, αν θέλετε, ε, πρόμηση, διότι έχουμε ήδη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, με σαφή προσανατολισμό προς την προώθηση του θέματος, αναφέρθηκε προηγουμένως η Επίτροπος, και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι και στον ευρωπαϊκό και το διεθνή τύπο αναδεικνύεται αυτή η ανάγκη. Είπε μάλιστα η Επίτροπος προηγουμένως, ας τροφοδοτήσουμε και εμείς αυτό το κλίμα συζήτησης που έχει, έχει δημιουργηθεί, για να μην πέσει η δυναμική, αντιθέτως να αναδειχθεί και να, ενισχυθεί. Ε, στην έκθεση λοιπόν παίρνουμε σαφή θέση ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση με τις επιχειρήσεις, να καταλάβουν την πρόκληση. Δεν αρκεί να προβάλλουμε κάποια παραδείγματα θετικά κάποιων επιχειρήσεων. Η Deutsche ε, Telekom και, και άλλες επιχειρήσεις έχουν σαφή καλές εμπειρίες να αναδείξουν. Πρέπει αυτό να γίνει μια γενική πρακτική. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε με τις επιχειρήσεις, να καταλάβουν την υποχρέωσή τους, ε, να καταλάβουν το το συμφέρον τους. Αναλύεται στην έκθεσή μου πώς αυτό συμβάλλει η συμμετοχή των γυναικών. Έχει σαφή αποτελέσματα, όλες οι έρευνες μας το δείχνουν. Όλα τα οικονομικά φόρα που γίνονται καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες είναι εξαιρετικές ε, ε, ε, και managers και administrators και πολύ, έχουν πολύ θετική έτσι, συμβολή διότι έχουν τα προσόντα, τα παιδείας και εκπαίδευση, είναι υψηλό το ποσοστό ε, παιδείας και εκπαίδευσης των γυναικών έχουν ε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συνένεσης, της προσοχής σε πολλές λεπτομέρειες, της αναζήτησης της καινοτομίας, του καινούριου, της προσέγγισης ε, της ποικιλομορφίας στο ανθρώπινο δυναμικό, στο δυναμικό της κοινωνίας. Πολλά χαρίσματα που έχει ανάγκη σήμερα η, η ευρωπαϊκή οικονομία για να ανταγωνιστής στο διεθνές και σκληρό επίπεδο. Λοιπόν, πρέπει οι να το καταλάβουν, να πάρουν ένα, μια σωστή κατεύθυνση ε, με ε, ε, προγράμματα αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Σε περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρουν, ε, ε, προτείνουμε να υπάρχουν πρωτοβουλίες, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με πρωτοβουλίες συγκεκριμένες το πώς θα θέσουμε στόχους δεσμευτικούς και μετρήσιμους. Αυτό είναι μια γενική προσέγγιση που πρέπει να ισχύει για όλους. Απ' την άλλη μεριά αναγνωρίζουμε μέσα στην έκθεση ότι η ευρωπαϊκή και κοινωνιακή οικονομία δεν είναι ομοιόμορφη. Ε, όπως και η κουλτούρα των επιχειρήσεων, ανάλογα με τη χώρα, με, τα θέμα, με το αντικείμενό τους δεν είναι ομοιόμορφοι. Υπάρχουν επιχειρήσεις που υπάρχουν πολλές γυναίκες ε, σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχουν επιχειρήσεις ε, που το αντικείμενο είναι τέτοιο που ε, βρίσκεται στη σφαίρα της ανδροκρατούμενης οικονομίας. Και υπάρχουν, όπως ας πούμε, οι μεταφορές, οι κατασκευές και υπάρχουν λιγότερες γυναίκες. Χρειάζεται λοιπόν ειδικέ προσεγγίσεις και μεθοδολογία για την κάθε περίπτωση, όπως και υπάρχει, και υπάρχει διαφορετική νομική κουλτούρα, ε, νομικό καθεστώς συγγνώμη, και ε, κουλτούρα διάρθρωσης των επιχειρήσεων. Άλλα όργανα έχει μια επιχείρηση διευθυντικά σε μια χώρα, αλλά υπάρχουν σε μια άλλη χώρα. Όλα αυτά θα τα λάβουμε υπόψη μας και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια αποφασιστική μετρήσιμη αλλά ήπια προσαρμογή για να πετύχουμε τους στόχους του 40% στα διοικητικά συμβούλια των γυναικών. Δεν έχει να κάνει την ίδια προσπάθεια μια χώρα που έχει 20% σήμερα και μια χώρα που έχει 6, που έχει 10. Σαφώς ε, πρέπει να υπάρχει μια αντιμετώπιση της ε, ε, ποικιλομορφίας που έχουμε σήμερα στην επιχείρηση. Άλλη ε, παρέμβασή μας έχει να κάνει με το ότι όταν ε, σχεδιάζουμε αυτή την έκθεση και αυτή την πολιτική παρέμβαση, στόχος μας δεν είναι μόνο να βρεθούν γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, στόχος μας είναι να βρεθούν γυναίκες που θεωρείται για αυτές, που καταλήγουν στα διοικητικά συμβούλια ως εξέλιξη της πορείας τους και της καριέρας τους μέσα στην επιχείρηση. Δεν θέλουμε δηλαδή με πρόσχημα το να βρεθούν γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, να δώσουμε την, ε, ε, το έναυσμα και το άλοφι στις επιχειρήσεις, να παίρνουν γυναίκες ε, από διάφορους χώρους, οι οποίες συνήθως έχουν και ένα επικοινωνιακό προφίλ, να τις τοποθετούν σε διοικητικά συμβούλια. Πολλές γυναίκες από την αγορά, από τη δημόσια ζωή, θα ήταν ωφέλιμες σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Στόχος μας είναι να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να επιδιώξουν μια δυναμική καριέρα και να έχουν την αναγνώριση τους ε, καταλήγοντας στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει παράλληλα να πάρουμε μέτρα, να πάρουν και επιχειρήσεις μέτρα για την ε, εξέλιξη των γυναικών σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης. Οι γυναίκες που θα είναι πιθανές καλές ε, ε, Καλά μέλη διοικητικών συμβουλίων είναι οι γυναίκες οι οποίες είχαν την ευκαιρία να έχουν θέσεις ευθύνη σε διάφορα επίπεδα της επιχείρησης. Άρα χρειάζεται μια υποστηρικτική προσπάθεια και πολιτική σε όλα τα επίπεδα. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να συνδυαστεί με την προσπάθειά μας είναι να, να, να υπάρξει μια κουλτούρα ε, αντισυσσόρευσης πόστων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν, ε, παραδείγματο χάρη, ε, και άνδρες και γυναίκες που λόγω ικανότητα πείρας έχουν, βρίσκονται σε δέκα διοικητικά συμβούλια. Νομίζω ότι και η αποτελεσματικότητα δεν συνάδει με την ε, συσσόρευση αρμοδιοτήτων ε, και από την άλλη πλευρά εμποδίζει το να υπάρχουν θέσεις ελεύθερες που θα μπορούσε, για τις οποίες θα μπορούσε να είναι υποψήφιες οι γυναίκες. Θέλω να πω κυρία Πρόεδρε και θα σταματήσω εδώ ότι ο στόχος μας είναι σαφής, η προσέγγιση μας είναι ρεαλιστική, ισορροπημένη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις που υπάρχουν σήμερα σε όλα τα επίπεδα, αλλά και η προσέγγιση μας είναι επίσης σφαιρική. Χρειάζονται πολλές ενέργειες παράλληλα, μέσα στην επιχείρηση, έξω από την επιχείρηση, ε, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο και να είναι το αποτέλεσμα μιας δυναμικής καριέρας των γυναικών που έχουν τα προσόντα και που θέλουν να παίξουν ρόλο στα ανώτατα επίπεδα διαχείρισης και αποφάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα θερμό ευχαριστώ, κυρία Κράτσα. Η κυρία Κώστα θα πάρει το λόγο, παρακαλώ. Συγγνώμη γιατί θα χρειαστεί να φύγω αμέσως, αλλά ήθελα πραγματικά να τοποθετηθώ στην έκθεση της συναδέλφου Κράτσα που είναι πάρα πολύ καλή και συμμερίζομαι αυτό το οποίο λέει ότι το θέμα των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά δεν θα πρέπει να αποτελέσει άλοθη για τις επιχειρήσεις για την πρόθεση των γυναικείων σταδιοδρομιών και η εμπειρία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σαφώς πιο συμβατή με αυτό το οποίο είπατε. Σε αυτή, την έκθεση διαπιστώνουμε πολλά στοιχεία της corporate governance και στην ε- ΕΚΟ και στην ΙΝΚΟ αλλά και στην Κομισιόν την ίδια η οποία το ψάχνει το θέμα. και η τροπολογία η σχετική με την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων ε, δεν θα πρέπει να ε, αποτύχει γιατί η τροπολογία δεν είχε περάσει για μία ψήφο. Ελπίζω να περάσει λοιπόν από τις άλλες επιτροπές. Ένα από τα εμπόδια για τις ε, γυναίκες ε, ως μάνατζερ είναι το θέμα των ε, δυσκολιών, δηλαδή ως εργαζόμενες ή ως επιχειρηματίες και θα πρέπει να επιμείνουμε για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και να υπάρχει κιόλας και ένα ευρωπαϊκό σήμα το οποίο να αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν αναλάβει ε, ε, δικό τους τον κώδικα της ηθικής ευθύνης ε, της επιχείρησης. Για παράδειγμα να είναι μια family friendly επιχείρηση ή να ενισχύει τη συνεχή κατάρτιση των γυναικών ούτως ώστε αυτές να καταφέρνουν να παίρνουν διευθυντικές θέσεις. Πρέπει επίσης ε, να ε, επεκτείνουμε το ζήτημα και στην ε, κοινωνική οικονομία. Μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ενώσεις όπου οι γυναίκες είναι παρούσες και όπου πρέπει να ενισχύσουμε την ανάληψη διευθυντικών ρόλων. Επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί η ανάγκη των γυναικών μάνατζερ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των μίντια. Διότι εμείς ε, σήμερα πρέπει να ντρεπόμαστε για το ρόλο των γυναικών σε όλα αυτά τα δημιουργικά μέσα επικοινωνίας και τη διαφήμιση. Και το τοπίο έχει αρχίσει και γίνεται γκροτέσκο κυρίως στην Ιταλία όσον αφορά στις ε, διευθυντικές ε, θέσεις ε, των γυναικών στα ΜΜΕ. Επίσης, θα πρέπει να καλέσουμε τις περιφέρειες που χρησιμοποιούν κονδύλια του κοινωνικού ταμείου να τα χρησιμοποιήσουν για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών και της παρουσίας τους στις διευθύνσεις επιχειρήσεων και αυτό και για τις μετανάστριες πρέπει να γίνει αυτό και στο πλαίσιο της έκθεσής σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κώστα. Η κυρία Σέσκοβα είναι η επόμενη ομιλήτρια, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κράτσα για την έκθεσή της. Και έχω και εγώ ορισμένες στοιχεία που έχω δει σε επίπεδο στατιστικό και έχω συμπεράνει ότι στην Τσεχία, στη χώρα μου, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις εξουσίας σε επιχειρήσεις είναι μονάχα το 9,5%. Είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό αυτό και είμαι προσωπικά πεπισμένη ότι ο κύριος λόγος γι' αυτό είναι τα παλαιά τετριμένα στερεότυπα, ότι η γυναίκα πρέπει να είναι στο σπίτι και να προσέχει τα παιδιά. Ένα παράδειγμα. Χθες σε ένα φόρουμ στο διαδίκτυο γινόταν μια συζήτηση και κάποιος έκανε μια δήλωση λέγοντας πώς μπορώ εγώ να είμαι ευρωβουλευτής χωρίς να έχω παιδιά. Αυτό είναι στερεότυπο. Αυτά τα στερεότυπα στα οποία αναφέρομαι. Τέτοια στερεότυπα οδηγούν κατευθείαν σε περαιτέρω συνέπειες και μία από τις σημαντικότερες συνέπειες και αυτό αφορά πάρα πολλές γυναίκες σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Μία από τις σημαντικότερες ε, συνέπειες μιας τέτοιας λογικής είναι ότι οι άνδρες έχουν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στην εργασία τους ως ανώτερα στελέχη και μπορεί ένα άντρα να εργάζεται νύχθη μερών ω τέλο, κάτι που δεν μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Αυτή λοιπόν είναι η προσέγγιση μου και εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα, ο πυρήνα του προβλήματο βρίσκεται σε αυτά τα στερεότυπα. Για το σχέδιο έκθεση τώρα, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Κράτσα για το σχέδιο έκθεσής της και θα ήθελα να σταθώ τώρα στο σημείο 3 Πιστεύω ότι εδώ αυτό μπορεί να είναι ένα επίμαχο σημείο. Γνωρίζω από την ίδια μου την εμπειρία ότι οι άνδρες πολύ συχνά έχουν θέσεις σε διοικητικά συμβούλια μονάχα για λόγους τιμής και για λόγους ε, κύρους και προβολής. και υπάρχουν αυτές οι θέσεις οι οποίες για μένα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στο σημείο 4 επίσης τονίζεται η σημασία του να υπάρχει και κάποια δυνατότητα συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Εδώ όμως θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο μήπως θα πρέπει να τονίσουμε περαιτέρω και το σημείο ότι το πιο σημαντικό σε αυτό το τομέα είναι η φροντίδα των πολύ νεαρών παιδιών. Θα πρέπει εδώ να κάνουμε λοιπόν τις απαραίτητες ενέργειες, να μπορούν οι εταιρείε να έχουν παιδικούς σταθμούς και να υποστηρίζουν τους παιδικούς σταθμούς, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να υποστηρίξει τους ε, γονείς αυτών των παιδιών, οι οποίοι θα πρέπει να εργάζονται μακρές ώρες και αυτό ισχύει ιδίω για τα υψηλά στελέχη. Και θέλω να έρθω και στο σημείο 7 επίσης, που αφορά <clears throat> τις ε, ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν σε νομικό και οικονομικό επίπεδο στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα ήθελα το σημείο αυτό να το διευρύνει λιγάκι η και συγκεκριμένα. Πρόκειται για το εξή, το κάθε κράτος ε, μέλος φυσικά έχει το δικό του νομικό πλαίσιο που <clears throat> δεν είναι εναρμονισμένα αυτά τα πλαίσια μεταξύ τους. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες και διάφοροι κανόνες στο εργασιακό πλαίσιο. Στην τσεχική δημοκρατία, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε συμβούλια επιχειρήσεων ή σε εποπτικά συμβούλια, ακολουθούν μια συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, αλλά η οποία δεν είναι η ίδια σε όλα τα κατημέλια. Και εδώ θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει σαφήνεια κανόνων και ορισμών για τις επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι από τις επιχειρήσεις αυτές σε σχέση με την ισότητα, θα πρέπει να υπάρχει και σαφής ορισμός της νομικής μορφής αυτών των επιχειρήσεων, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζεται σωστά μέσα στην ένωμη τάξη του κάθε κράτους. Οι στρατηγικοί που έχουμε δείχνουν ότι μπορούν να υπάρχουν πολλαπλά ε, κριτήρια για τις επιχειρήσεις αυτές ανεκ σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Ίσως οι σκιώδεις εισηγητές μπορούν να διεξέλθουν το θέμα αυτό όταν συζητήσουν με την κυρία εισηγήτρια για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιους κανόνες οι οποίοι μπορεί να είναι εναρμονισμένοι αλλά μπορεί να είναι και σαφείς και να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες ώστε να μπορούμε να ξέρουμε τι λέμε όταν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ποσοστό γυναικών σε υψηλέ θέσεις. Ευχαριστώ, λέει και Η κυρία Ουβίρ τώρα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την έκθεση της κυρίας Κράτσα. Μελέτησα πολλές φορές εις βάθος ε, την έκθεση αυτή. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσθέσω οτιδήποτε, διότι είναι πληρέστατη η έκθεση και ε, καλύπτει το σύνολο των πτυχών του ζητήματος. Ε, πρόσφατα στον Ταβός, στην συνεδρίαση των ηγετών του επιχειρηματικού κόσμου, ε, οι εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρήσεων, των πλέον καινοτόμων επιχειρήσεων, έκαναν κάποιες δηλώσεις που συνάδουν με το περιεχόμενο της έκθεσης. Ε, ε, αυτό είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο για την υλοποίηση των στόχων της έκθεσης συγκεκριμένα για να μετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Η πολιτική ελίτ τώρα, οι κυβερνήσεις, ποια στάση έχουν τηρήσει. Στην πατρίδα μου πριν από μία εβδομάδα είχαμε εκλογές. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την οικοδόμηση κυβέρνησης συνασπισμού. και ε, ε, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τουλάχιστον δύο γυναίκες υπουργούς για να φτάσουμε το ποσοστό του 10% για τη συμμετοχή των γυναικών. Το Υπουργείο Πολιτισμού ελπίζουμε να έχει επικεφαλής μία γυναίκα γιατί δεν υπάρχουν μόνο τα οικονομικά προβλήματα σε μία κοινωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ορισμένες ε, χώρες να υλοποιηθούν οι εξαιρετικές ιδέες αυτής της έκθεσης λόγω της πολιτικής κατάστασης. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θα μπορούσε η συγγήτρια να τονίσει και κάποια, τη σημασία κάποιων νομικών ρητρών που θα ε, επέβαλαν στα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τις δράσεις και τις ιδέες της έκθεσης. Πάντως ε, ε, χαίρομαι που είναι σαφέστατη η πολιτική θέση που τηρεί το Κοινοβούλιο για το ζήτημα αυτό. Οι ποσοστώσεις ε, δεν είναι όπως γνωρίζουμε το βασικότερο εργαλείο ελοπίστων των στόχων μας, υπάρχουν και άλλα πολλά μέσα, άλλα πολλά εργαλεία που μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν. Η αποκλειστική χρήση των ποσοστώσεων ε, δεν επαρκεί σε κάποιες κοινωνίες και πάλι. Να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια και να ευελπιστώ ότι θα υπερψηφιστεί η έκθεση. Ευχαριστούμε η κυρία Μπάστους τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την ε, κυρία Κράτσα και κατά δεύτερο λόγο να διαβάσω ένα μήνυμα που μου άφησε η κυρία Μωράν Σαρτιέ για να διαβιβάσω εξ ονοματός της σε σχέση με την έκθεση αυτή δεδομένου ότι η Ελιζαμπέτα δεν μπορεί να είναι παρούσα γιατί έχει μια άλλη συνεδρία σε μια άλλη συνεδρίαση. Θα ήθελα να πω στην κυρία Ρόδη Κράτσα ότι έχει κάνει ένα πάρα πολύ σωστό ε, έχει πάρει μια πολύ σωστή τοποθέτηση για το θέμα αυτό και την κατάσταση των γυναικών στα, στους φορείς λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και βλέπω ότι αντιμετωπίζει πράγματι το πρόβλημα να υπάρξει μια αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στους φορείς λήψης απόφασης. Η λύση αυτού του προβλήματος περνάει από κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι και τονίστηκε πολύ σωστά από την εισηγήτρια και από άλλες <clears throat> συναδέλφους, το να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τα μέτρα τα οποία συμφιλειώνουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητο χώρο στι γυναίκε με προσόντα για να μπορέσουν αφενό να συνεχίσουν τι καριέρε του και συγχρόνω να διατηρούν την οικογενειακή του ζωή. Θα ήθελα επίση για όλα αυτά που είπε η συγγήτρια να πω ότι είναι απόλυτα λογικά και τεκμηριωμένα αυτά τα οποία προτείνει και συνάδουν με αυτά που τόνισε και η ίδια η Επίτροπος ε, Ρέδιν ότι θα πρέπει από την πρώτη στιγμή να ζητήσουμε την ε, υποστήριξη του χώρου των επιχειρήσεων ώστε να υπάρξουν οι βέλτιστες πρακτικές για να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια οι γυναίκες και αυτά μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ λογικά, ότι είναι μέτρα τα οποία έλκονται και από την κοινή λογική. Και επίσης το ερώτημα του αν μόνο με βέλτιστες πρακτικές και εθελοντικές ε, κινήσεις των επιχειρήσεων αν δεν μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, τότε σε τελική ανάλυση για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι θα πρέπει προσωρινά και εκτάκτως να καταφύγουμε σε ποσοστώσεις. Νομίζω ότι η κυρία Κράτσα το θέτει αυτό το θέμα με μεγάλη σαφήνεια. Και τώρα θα σας διαβάσω το μήνυμα της κυρίας Μωρέν Σάρτιε. Σας δίνω όλη την υποστήριξή μου στο σχέδιο της κυρίας ε, Κράτσα και την εξαιρετική της δουλειά που θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στις εξελίξεις, στις απαραίτητες εξελίξεις που πρέπει να αναλυθούν στα διάφορα σημεία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επενδύσουν στην κατάρτιση των νέων γυναικών και των οποίων όμως η κατάρτιση δεν ανταποκρίνεται. Θα πρέπει να τους δοθεί λοιπόν κατάρτιση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν με το 100% της ευθεία τους ε, και με το φιλεργατικό τους αίσθημα. Σε μία περίοδο κρίσης θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια ούτως ώστε οι γυναίκες να μπορούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνες. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις οι οποίες άσκησαν πολιτικές ισότητας μεταξύ ανδρών γυναικών και που υποστήριξαν την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ε, ε, διευθυνσής άντεξαν καλύτερα την οικονομική κρίση. αυτή τη δυναμική αυτή η δυναμική είναι η σωστή δυναμική για την απασχόληση και πρέπει να την αναπτύξουμε. Έχουμε να κερδίσουμε τα πάντα. Τρίτο, συμφωνώ απόλυτα στις προτάσεις ε, της ε, κυρίας ε, Κράτσας. Κράτσα, θα ήθελα ε, οι γυναίκες να μπορέσουν να αναγνωριστούν στην εργασία τους και αυτό στη βάση των ικανοτήτων τους. Πρέπει όμως να παραδεχτώ ότι αν δεν ορίσουμε και με στόχους που μπορούμε να τους μετρήσουμε μέσα στις επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εξέλιξη των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τις προτάσεις της και επίσης λέω ότι πρέπει να πάμε προς την ίδια κατεύθυνση και στο δημόσιο τομέα. Η κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμμερίζομαι και υποστηρίζω όλα τα κίνητρα που έσπρωξαν την κυρία Κράτσα να συντάξει αυτή την έκθεση, μία εξαιρετική έκθεση η οποία βρίσκεται στην καρδιά της επικαιρότητα. Στην καρδιά της επικαιρότητα όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ορισμένων κρατών μελών μεταξύ των οποίων και της Ιταλίας που ψηφίζει σήμερα στην Γερουσία τον νόμο για την ποσόστοση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Ρωτώ την κυρία Κράτσα, μήπως θα έπρεπε να εγκρίνουμε και πολιτικές ad hoc έναντι των επιχειρήσεων εκείνων που θα δεχθούν να συμμετέχουν και να εφαρμόσουν αυτήν την μελλοντική ευρωπαϊκή οδηγία. Να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτές τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την πολιτική ε, γυναικών στελεχών να υποστηρίξουν και την κοινωνική πολιτική υπέρ της οικογένειας. Να υποστηρίξουμε επίσης και πιλωτικά σχέδια, ούτω ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για το σωστό συνδυασμό μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Σας ευχαριστούμε. Τώρα είναι η δική μου σειρά. Θα ήθελα να αναφέρω ότι είμαι κι εγώ σκιώδης εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε κυρία Κράτσα. Ε, κατά τη γνώμη μου είναι ορθότατο και πληρέστατο το περιεχόμενο της έκθεσης. και ως σκιώδης εισηγήτρια ακόμη δεν κατάφερα να εντοπίσω ποια σημεία θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε μέσα στην έκθεση. Ήδη υπάρχουν, ε, καλύπτονται σχεδόν όλες οι πτυχές ε, του ζητήματος. Θα δούμε σε μελλοντική εξέταση της έκθεσης αν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Συγχαρητήρια κυρία Κράτσα ε, για την έκθεσή σας είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά επίκαιρο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και γεννά μεγάλη δέσμευση και έντονο διάλογο σε όλα τα κράτη-μέλη. Με αυτήν την συζήτηση αυξάνουμε την επίγνωση για αυτό το ζήτημα και άλλα ζητήματα ισότητας των δύο φύλων και έτσι μπορούμε να δώσουμε καλύτερες ευκαιρίες στις γυναίκες να αξιοποιηθούν τα προσόντα τους, όπως πολύ σωστά αναφέρετε στην έκθεσή σας. Επιχειρηματολογούμε στα πλαίσια αυτής της συζήτησης, ε, χρησιμοποιώντας ε, οικονομικά στοιχεία επίσης, ότι είναι δηλαδή επικερδές για την ίδια την επιχείρηση όταν συμμετέχουν πολλές γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε διευθυντικές ε, θέσεις. Αυτό το επιχείρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όντως χρειαζόμαστε τα προσόντα και τις εμπειρίες των γυναικών στην επιχείρηση και από οικονομικής πλευράς είναι θετική συμμετοχή τους. Έχει ιδιαίτερο βάρος αυτό το επιχείρημα. Για μένα όμως υπάρχει και ένα άλλο εξίσου σημαντικό. Η ισότητα των δύο φίλων στο εσωτερικό μίας επιχείρησης είναι αυτό καθεαυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η ισότητα είναι ένα ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Οι άντρες και οι γυναίκες δικαιούνται ε, ισότιμη μεταχείριση. Οπότε θα μπορούσαμε ε, σε αυτή την συζήτηση να καταδείξουμε με συγκεκριμένα στοιχεία πόσο θετικό από οικονομικής πλευράς είναι για την επιχείρηση να συμμετέχουν οι γυναίκες. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, συχνά συζητούμε το θέμα των στερεοτύπων των δύο φύλων, ότι βάζουμε δηλαδή τους άντρες και τις γυναίκες σε διαφορετικά καλάθια και οι διευθυντικές σχέσεις επιχείρησης ε, ε, στελεχώνονται από το καλάθι των αντρών. Είναι ένα συχνό στερεότυπο. Εμείς θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτό το στερεότυπο και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το επιχείρημα. Στο σημείο 3 της έκθεσης ε, κάποιος αναφέρθηκε σε αυτό. Εκεί η συγγήτριά μας, η κυρία Κράτσα, ε, αναφέρει ε, ότι ε, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε την σημασία το, του ρόλου των γυναικών στις διευθυντικές ε, θέσεις και θεωρώ ότι όπως ε, σωστά είπατε δεν θα πρέπει να παραχωρούνται τέτοιες θέσεις στα διευθυντικά όργανα σε γυναίκες τιμής ένεκεν αλλά μόνο σε γυναίκες που έχουν αποδείξει την αξία τους εντός των επιχειρήσεων υποστηρίζω πλήρως αυτό το σημείο και θα κλείσω ένα λεπτάκι μόνο για τις ποσοστώσεις ε, ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά Χρειάζεται αυτό το εργαλείο, είναι απαραίτητο για να καταφέρουμε να αλλάξουμε την ε, κατάσταση. Δεν, ε, χρησιμοποιεί, δεν ε, λειτουργεί σωστά το σύστημα όταν 97% των διευθυντικών θέσεων στις μεγάλες επιχειρήσεις έχουν καταληφθεί από άντρες, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν είναι σωστό, κάτι έχουμε κάνει λάθος. Δηλαδή μόνο 3% γυναικών έχουν τα πετούμενα προσόντα για να καταλάβουν αυτά τα αξιώματα στις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να αληθεύει αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία του εργαλείου των ποσοστώσεων στον αγώνα που θα δώσουμε. Υποστηρίζω λοιπόν την προσέγγιση της Κυρία Κράτσα. Προφανέστατα η επιχείρηση μέσω της διαδικασίας αυτορύθμισης θα πρέπει να επιληθεί του ζητήματο Συμφωνώ, αλλά σε έχουμε και πλήρη επίγνωση του ότι αν δεν λειτουργήσει η αυτορύθμιση τότε θα πρέπει να παρέμβουμε με το σύστημα των ποσοστώσεων ε, στις επιχειρήσεις. Εξαιρετική η έκθεσή σα, κυρία Κράτσα και θα κλείσω εδώ δίνοντα ε, το λόγο στην κυρία Βέρτμαν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Και από αυτά που άκουσα βλέπω ότι η Τσεχία και η Αυστρία έχουν παρόμοια προβλήματα. Και εγώ άκουσα ότι στη δική μου εκλογική εκστρατεία ότι θα πρέπει και εγώ να έχω να ασχολούμαι περισσότερο με τα μητρικά μου καθήκοντα. Βέβαια, η κόρη μου είναι αρκετά μεγάλη και δεν έχει πρόβλημα με αυτά τα οποία κάνω. Υπάρχουν και στην Αυστρία πάρα πολύ έντονα προβλήματα και προκαταλήψεις. Λένε ότι η γυναίκα θα πρέπει να μείνει στην κουζίνα και να φροντίσει τα παιδιά της. Λένε πολλές φορές ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν τα ίδια προσόντα αλλά και οι άνδρες δεν έχουν πολλές φορές τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα ίδια πράγματα τα οποία κάνουν οι γυναίκες. Λοιπόν, ήδη θα πρέπει και οι άνδρες να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους στο να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του οίκου. Οι γυναίκες δεν έχουν χαμηλότερα προσόντα σε επιχειρήσεις από ότι οι άνδρες. Όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Ρέντινγκ, και νομίζω ότι οι ποσοστώσει θα πρέπει να είναι απλώ ένα βοηθητικό εργαλείο μέχρι το σημείο που θα μπορέσουμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια ισορροπία 50-50% και η ισορροπία στον τομέα αυτό και στο σημείο τώρα 3 εγώ θα ήθελα να προσθεθεί το γεγονός ότι υπάρχουν και γυναίκες έξω από μια επιχείρηση οι οποίες λόγω της γνώσης τους και των προσώπων τους μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση και επίσης το σημείο 4 που έχει να κάνει με, την, με τη συμφιλίωση της εργασιακής και της ε, οικογενειακής ζωής θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπε η κυρία Ματέρα για να δοθούν και φορολογικά κίνητρα. Νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε τέτοια κίνητρα από την πλευρά των, ε, για τις επιχειρήσεις ώστε να έχουν φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, κάτι το οποίο θα δώσει δυνατότητα στους ε, εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε επίπεδο υψηλό στην επιχείρηση να έχουν την φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων γονέων τους χωρίς να αφαιρούν χρόνο από τον χώρο εργασίας. Θα ήταν αυτό παραπολυθετικό για να εξασφαλίσουμε μια ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν εξάλλου πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ ψηλά προσόντα, αλλά παίρνουν σημαντικά λιγότερα χρήματα από άνδρες εργαζόμενους. Επομένως, η ισότητα σημαίνει για την ίδια εργασία και ίδια <clears throat> αμοιβή και για τα ίδια προσόντα επίσης να υπάρχει η διαμοιβή. Εδώ στην χώρα μου πολλές φορές γυναίκες με υψηλότερα προσόντα παίρνουν πολύ λιγότερα ε, λεφτά από άνδρες με λιγότερα προσόντα. Σας ευχαριστούμε και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζαμπόσκα, παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εξάρω το έργο της κυρίας Κράτσα. Είναι πολύ καλή και ισορροπημένη η έκθεσή της. Προσπάθησε να καλύψει το πλήρες φάσμα προβληματικής για τα θέματα αυτά και ξέρουμε φυσικά ότι είναι πολλαπλά τα θέματα τα οποία γύρονται σε σχέση με την ισότητα μεταχείριση. Εγώ θέλω να σταθώ μονάχα σε ένα σημείο το οποίο αναφέρει η κυρία Κράτσα και στην έκθεσή τη. Πρόκειται για το εξή σημείο. Όταν εμεί δεν δίνουμε δυνατότητα στου άνδρε αλλά και στι γυναίκε να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή, αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία μας σπαταλάει το ταλέντο και τις δυνατότητες ανθρώπων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να επιλύσουμε αυτό το πολύπλοκο πρόβλημα και να δώσουμε τις δυνατότητες και στις γυναίκες να μπορούν να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας μας. Και θέλω να σας υπενθυμίσω αυτά τα οποία είπε η κυρία Ρέντινγκ προηγουμένως. Τα λέει και η κυρία Κράτσα στην εκθεσή της και καταδεικνύει την κατάσταση σε ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία, κάτω χώρες Βέλγιο και Γερμανία. Πρόκειται για χώρες οι οποίες έχουν προσπαθήσει να επιτύχουν με ποσοστώσεις και άλλα μέτρα την ε, ανύψωση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ε, ε, ευθύνης. Και αν δούμε τώρα τις προθεσμίες οι οποίες προβλέπονται για την επίτευξη αυτών των στόχων βρίσκονται στο, στο, στον ορίζοντα του 2014-2015. Αν επιτευχθούν όλα αυτά θα είναι πολύ θετικό. Παραδέχτηκε η κυρία Ρέντινγκ ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εφικτό μέχρι το 2012 να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη ισο εκπροσώπηση των γυναικών. Αλλά τόνισε ότι αν δεν επιτευχθεί αυτό μέχρι το 2012 θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε νομοθετικά μέτρα. Εγώ όμω πιστεύω ότι είναι καλύτερο αντί να ρυθμιστεί αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο το κάθε κράτο μέλος να ακολουθήσει τη δική, της, τη δική του οδό γιατί αλλιώ θα έχουμε πολύ μεγάλε αντιδράσει. Αυτό θα ήταν κρίμα. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε για τα θέματα αυτά για να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το φράγμα το οποίο εμποδίζει τις γυναίκες εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι αυτά τα οποία προτείνουν τα την κυρία Κράτσα στο σημείο 4 για τα μέτρα τα οποία πρέπει να αναλυφθούν θα συμβάλλουν τα μάλα για τη βελτίωση της κατάστασης και για να μπορέσουν οι γυναίκες να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και να είναι καλύτερα εκπροσωπούμενες στα ανώτερα κλιμάκια των επιχειρήσεων εγώ νομίζω ότι η κυρία Κράτς έχει αντιμετωπίσει πολύ σωστά αυτό το πολύπλοκο θέμα και αξίζει κάθε υποστήριξη η έκθεσή της. Σας ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα τον, ε, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώ συγγνώμη. Thank you very much, Madam Chair. And, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, γνωρίζετε την δέσμευση και την αφοσίωση της Επιτρόπου Ρέντινγκ για αυτό το θέμα. Επίσης γνωρίζετε ότι υπάρχει μια νέα στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων που έχει ήδη εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλωσορίζουμε την έκθεση που προετοιμάζεται στην Επιτροπή σας. Θα θέλαμε μόνο να υπενθυμίσουμε τα εξής το παρελθόν αλλά και τώρα. Υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ άλλων και με χρηματοδοτικά μέσα, ε, τα προγράμματα και τις δράσεις των διαρθρωτικών ταμείων για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επί σειρά ετών ε, χρηματοδοτήσαμε εκστρατείες ενημέρωσης ε, στα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και γενικότερα τα διαρθρωτικά τα μία ε, έχουν, όπως γνωρίζουν οι αξιότιμοι βουλευτές, ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να ενισχύσουν το ρόλο των γυναικών ως προς τη λήψη αποφάσεων. Ε, να σας υπενθυμίσω επίσης κάτι για τη βάση δεδομένων για τις γυναίκες και τη λήψη αποφάσεων. Σήμερα συζητούμε για τους στόχους και τις ποσοστώσεις. Πρέπει να ε, μετράτε η πρόοδος που σημειώνεται για την επίτευξη των στόχων. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων λοιπόν για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Επίσης, ετησίως υποβάλλουμε μία έκθεση προσκομίζοντας τα στοιχεία ε, που έχουμε συλλέξει στη βάση δεδομένων και όπως γνωρίζετε εκδώσαμε μόλις μία έκθεση για ε, την ισότητα των δύο ε, φύλων τη διεύθυνση των επιχειρήσεων. Έχετε αντίτυπα, αν θέλετε, βγαίνοντα από την αίθουσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε, κυρία Τομασέτη. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην ε, κυρία Κράτσα για να κάνει τα καταληκτικά της σχόλια. Παρακαλούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, είμαι με πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Άκουσα τα σχόλιά σας και θεωρώ μια πολύ καλή προοπτική για την τελική έκβαση το ότι συμμεριζόμαστε και τις γενικές ε, κατευθύ... το στόχο αυτής της έκθεσης αλλά και τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προτείνονται. Ε, καταρχάς για τις παρατηρήσεις της κυρίας Κώστα, έστω και αν δεν είναι εδώ η κυρία Κώστα, ήθελα να διευκρινίσω ότι το πεδίο εφαρμογής είναι οι γυναίκες στα διευθυντικέ στις διευθυντικές θέσεις των επιχειρήσεων και όχι οι γυναίκες επιχειρηματίες. Το λέω αυτό γιατί η κυρία Κώστα έκανε αναφορά σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, αλλά δεν αποτελεί το αντικείμενο της έκθεσης, που είναι οι γυναίκες που έχουν τη δική τους επιχείρηση και πόσο σημαντικών για την οικονομία και την κοινωνία. Θεωρώ πολύ σημαντική την παρατήρηση της κυρίας Κώστα ότι αυτή η προβληματική που αναπτύσσεται δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις που ομολογουμένως ήταν και είναι και το πεδίο της εφαρμογής στη δική μου σκέψη αλλά και στην κοινωνική οικονομία. Ε, πολλές μικρές επιχειρήσεις, πολλές ε, επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα και σε αυτές πρέπει να υπάρχει αυτή η, αν όχι δέσμευση σε αυτή την περίπτωση, αλλά η πολιτική και η νοοτροπία της ίσης εκπροσώπησης. Ε, η κυρία Σέσκοβα αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα άρθρα μάλιστα, το άρθρο 3 και το, και το σημείο 3 του άρθρου 4. Ως προς το άρθρο 3, νομίζω ότι η κυρία Σέσκοβα ήθελε να πει ότι ε, ε, τιμητικές θέσεις έχουν και άνδρες σε κάποια διοικητικά συμβούλια, γιατί να μην τα έχουν και κάποιες γυναίκες. Ε, φυσικά αυτό το αντιμετωπίζω με μια τροπολογία που έχω σκοπό να κάνω και ήδη σας αναφέρθηκα σε αυτό ότι δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συγκέντρωση ε, θέσεων στα διοικητικά συμβούλια πέντε άξιοι άνδρες και δύο άξιες γυναίκες μπορούν να έχουν 25 ε, θέσεις σε διοικητικά συμβούλια. Λοιπόν, ό,τι ισχύει για τους άνδρες ισχύει και για τις γυναίκες, αλλά νομίζω ότι το πνεύμα του άρθρου αυτού είναι να δώσει έμφαση όχι ότι ε, πρέπει να υποτιμούμε τις γυναίκες που κάνουν καριέρα στην επιχείρηση ή να μην έχουμε τη δυνατότητα να τις ανακαλύψουμε και να τις αξιοποιήσουμε. Ε, ε, σέβεται το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, ε, αν κατάλαβα καλά, ε, ίσως είναι σε άλλο, έχει κάνει άλλη σκέψη, εκτός περιεχομένου του άρθρου, κυρία Σέσκοβα. Επίσης θέλω να αναφερθώ στις άλλες παρατηρήσεις, κυρία Σέσκοβα. Πρώτον, ότι πρέπει ε, στο σημείο που λέμε τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς στις επιχειρήσεις, ότι πρέπει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Ε, ξέρετε, προσπάθησα μέσα σε νέα μόλις άρθρα να έχω μια ε, περιεκτική αντιμετώπιση του θέματος. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, υποστηρίζουμε τους στόχους της Βαρκελόνης όλοι ε, και δεν βλέπω ότι χρειάζεται να γίνει εδώ αναφορά στα μικρά παιδιά. κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ξέρει πού είναι οι ανάγκες των εργαζομένων και σαφώς οι ανάγκες στις, ε, στις μικρές ηλικίε είναι αυτονόητες. Δεν αισθάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα δώσει προστιθεμένη αξία αν το θίξουμε εδώ. Αναφέρθηκε επίσης η κυρία Σέσκοβα στο ότι υπάρχουν ε, δεσμεύσεις νομικές διαφορετικές, καθεστώτα διαφορετικά νομικά στις διάφορες χώρες. Νομίζω ότι σαφώς αυτό το αναφέρω στο σημείο Β του άρθρου 7 Λέω σαφώς ότι και η επικουρικότητα πρέπει να γίνει σεβαστή και οι, οι, διαφορετικές ε, ε, συνθήκες ή των δομών των επιχειρήσεων, των νομικών, ε, των νομικών επίσης δεσμεύσεων και αναφέρω και, το, και σε επίπεδο ε, περιφερειακό, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν περιφερειακές ιδιαιτερότητες, ε, δεν είναι μόνο οι ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Αν ε, νομίζει ότι είναι κάτι, κυρία Ζέσκοβα, κάτι άλλο το οποίο πρέπει να εντάξουμε που κάνει την ε, σκέψη αυτή πιο σαφή, είμαι στη διάθεσή σας. Ε, επίσης η κυρία Όβιρ, λείπει τώρα, <laughs> αναφέρθηκε στις νομικές ρήτρε, θα μπορούσε στο άρθρο 8, εκεί που λέμε ότι πρέπει να έχουμε ειδικέ και μετρήσιμες ε, ε, ε, δεσμεύσεις, να μπορούμε να συμπληρώσουμε νομοθετικές δεσμεύσεις. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα και ήδη είναι και στη δική μου σκέψη. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Μπάστος και την κυρία Μορέν, που παρόλο που δεν είναι εδώ μας σκέφτεται. Αυτό δείχνει πόσο κάνει ένα κονσένσους το θέμα αυτό μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας. Η κυρία Ματέρα αναφέρθηκε στην ε, ε, ανάγκη ε, του να υποστηριχθούν και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη διάθεση να συμβάλλουν στην άρση των εμποδίων. Ε, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ε, να κάνουμε μια παρένεση στα κράτη-μέλη αξιοποίησης όλων των εργαλείων των κοινοτικών, διότι τα διαρθρωτικά ταμεία ε, έχουν αυτό το στόχο να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν δράσεις υπέρ της ενίσχυσης της εισόδου και παραμονής στην αγορά εργασίας των γυναικών. Άρα έχουμε αυτά τα εργαλεία. Καλό είναι να τα προβάλλουμε περισσότερο για να μπορούν να τα κάνουν, να κάνουν και οι επιχειρήσεις ε, ε, χρήση. Επίσης, ήθελα να πω ότι και η κυρία Βέρτμον έκανε αξιόλογες ε, παρατηρήσεις ε, για το άρθρο 3, το οποίο περιμένω πώς θα διατυπώσει μια δική της σκέψη επ' αυτού. Ε, το άρθρο 3 βλέπω ότι έλκει την προσοχή πολλών συναδέλφων και επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη συμφιλίωσης. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι επειδή ασχολήθηκα διαβάζοντας πολλές μελέτες επί του θέματος αυτού, η βασική, από ό,τι φαίνεται, τίποτα δεν είναι ε, ε, απόλυτο, αλλά οι τάσεις μας λένε ότι το βασικό εμπόδιο δεν είναι η συμφιλίωση, ανέλυξη των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις, δεν είναι τόσο η διευκόλυνση ανατροφής των, των παιδιών και αντιμετώπιση οικογενειακών βαρών, όσο η κουλτούρα μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Δηλαδή το λέω αυτό διότι δεν πρέπει να ρίξουμε το βάρος σε αυτό το πρώτο εμπόδιο που μας έρχεται στο νου, που είναι η συμφιλίωση ε, ε, και ήδη που είναι κάτι χιλιοϊπωμένο και για το οποίο υπάρχουν και εργαλεία να αντιμετωπιστεί και εργαλεία κοινοτικά, αναφέρομαι πάλι στα διαρθρωτικά ταμεία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κουλτούρα που υπάρχει μέσα στην επιχείρηση και να δώσουμε και στις γυναίκες τις ίδιες την ευκαιρία και το έναυσμα να εκδηλώσουν τις φιλοδοξίες τους και να θελήσουν και οι ίδιες να παίξουν ένα ρόλο διευθυντικό. Επίσης πιστεύω ότι μια και βρισκόμαστε σε αυτή τη λογική της αντιμετώπισης του θέματος σε επίπεδο ευρωπαϊκό, πέρα από τις εθνικές προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και γι' αυτό όπως η κυρία Ζαμπόσκα είπε πολύ καλά, τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους και τις ευθύνες τους, διότι όταν δεν καταλάβουν την πρόκληση αυτή, με το ότι θα πάρουμε εμείς μια ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να έχει και αντιδράσει από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό χρειάζεται παράλληλα να κρατήσουμε το θέμα ζωντανό, όπως είπε και η Επίτροπος. Αυτό το διάστημα που δημιουργείται μια συγκυρία υπέρ της υπόθεσης αυτής, σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο ε, μέσω μαζικής ενημέρωσης, είναι καλό να γίνει μια ευρεία ενημέρωση. Ε, διότι έτσι και τα κράτη-μέλη θα καταλάβουν τις ευθύνες τους και οι ενέργειές θα είναι συμπληρωματικές με τις ευρωπαϊκές και οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα καταλάβουν το συμφέρον και τα περιθώρια που έχουν να δράσουν σε αυτόν τον τομέα. Και μια και βρισκόμαστε σε αυτή την υπόθεση, ήθελα να πω ότι πρέπει να δούμε και το θέμα ε, των ποσοστώσεων στα επίπεδα τα α, κοινοτικά των ευρωπαϊκών οργάνων. Ήδη υπήρχε μια τροπολογία για την, ε, ε, στην Ευρωπαϊκή, Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα έχουμε νέες υπηρεσίες ε, για τη ρύθμιση και την εποπτεία των, των αγορών. είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εντάξουμε και στη λογική την ευρωπαϊκή στα υπάρχοντα και στα νέα συμβούλια που δημιουργούνται διότι μόνο τότε θα πείσουμε και τα κράτη-μέλη ότι είναι ε, ε, σοβαρές ε, οι δεσμεύσεις που παίρνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν τις εφαρμόζουμε καταρχάς στα, όργανα τα οποία έχουν σχέση με, αμεσότερη με, με μας. Ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή που ήταν σήμερα παρούσα, ε, πέρα από τις δηλώσεις της Επιτρόπου και η εκπρόσωπος της Επιτροπής σήμερα που συνέβαλε ε, προς αυτή την ε, κατεύθυνση που παίρνει η, η έκθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ και πιστεύω ότι μετά από την πλούσια συζήτηση που έγινε ε, θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε κάποια πράγματα στην έκθεση για την αρτιότητα και την συμμετοχή και την ε, ανάληψη έτσι, της υποχρέωσης να συμπεριλάβει όλες τις απόψεις που ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το χρονοδιάγραμμα είναι 23 Μαρτίου μέχρι τις 12. Είναι η προθεσμία για την, την ε, υποβολή των τροπολογιών. Στις 20 Απριλίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια έχει προβλεφθεί ψηφοφορία για τον Ιούνιο. Φτάσαμε επιτέλους στο σημείο 16 τα διάφορα. Δεν έχουμε όμως κάποιο σημείο στα διάφορα. 17 τώρα, η ημερομηνία της προσεχούς συνεδριάσεως. 24 Μαρτίου θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση και κατόπιν στις 20 Απριλίου η κανονική τακτική μας συνεδρίαση. Είναι ώρα να κλείσουμε τη σημερινή μας ε, συνεδρίαση. Και κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια όλους τους ε, συναδέλφους στη Γραμματεία. Ευγενικά η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους ερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Ε, στο ε, επανειδής 24 Μαρτίου θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.